θα, θα μιλήσουν για τη Σύνοδο Κορυφής. Δεν θα ξεκινήσουμε λοιπόν στις 3 το απόγευμα, αλλά στις 4 παρατέταρτο. Έχουμε λοιπόν και την έκθεση Wilmot. Καλό θα είναι να έχουμε επαρκή χρόνο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Άρα παρακαλώ όλοι να είστε παρούσες και παρόντες στις 4 παρατέταρτο. Θα ψηφίσουμε και μετά θα προχωρήσουμε στη συζήτηση εκθέσεως Wilmot. Έχουμε όλες τις γλώσσες σήμερα εκτός των εσθονικών και των μαλτέζικων και στις 26 Μαρτίου στις 2 και 30 έως 5 και 30 προβλέπεται συζήτηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και παρακαλώ να συμμετάσχετε όσο το δυνατόν πολυαριθμότεροι. Και αύριο θα έχουμε και ομάδα επισκεπτών 18 επισκέπτες του κυρίου Σύρι Προβιέ από την Εστονία. Την 5η, 21 Μαρτίου, στις 11.30 έχει προσκαλέσει ομάδα επισκεπτών η κυρία Οκονή. Την προηγουμένη εβδομάδα διεξήχθη ο πρώτος τριμήρης διάλογος για το Stop the Clock με συγητή τον Πέτερ Λίζε και στον πρώτο αυτό διάλογο επιτεύχθηκε συμφωνία με το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα της οποίας θα ψηφίσουμε στις 26 Τρίτου. Και η τελική ψηφοφορία θα γίνει στην Ολομέλεια του Απριλίου. Χαίρο ιδιαίτερα που πήγαν τόσο καλά τα πράγματα για αυτή την τόσο σημαντική έκθεση, συν τόσο σημαντική αυτή νομοθετική διαδικασία. Έχουμε τα πρακτικά τώρα, 28-29 Νοεμβρίου, 18-19 Φεβρουαρίου και 28 Φεβρουαρίου. Αυτά προς ενημέρωση. Στο 4 διακόπτει ο Πρόεδρος. ω σας προσκαλούμε στην συνεδρία της Επιτροπής. Καλώς ήρθατε. πολύ ευχαρίστως να παραμείνετε. Έρχομαι, ερχόμαστε λοιπόν συγγνώμη, στον κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δώσω το λόγο για πέντε λεπτά στην εισηγήτρια και μετά θα αναγκαστώ βέβαια να σας περιορίσω σε δύο λεπτά μόνο, διότι έχω πολλούς εγγεγραμμένους και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλουμε επίσης να ακούσουμε και την Κομισιόν καθώς και άλλες παρεμβάσεις για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Άρα πρώτη η κυρία Ροτ Μπέρεν, στο μεταξύ σημειώνω ονόματα και θα κλείσω τον κατάλογο εν ευθέτω χρόνο. Η Ντάγμαρ, σε ευχαριστώ Ματίας. Λοιπόν πολύ τα έχω ετοιμάσει όλα στα αγγλικά. Και ο Νικολά εδώ, ο συνεργάτης μου, προτιμά τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Γι' αυτό το κείμενό μου θα είναι στα αγγλικά. Αν και συνήθως στην Επιτροπή δεν τα α, μιλώ τα αγγλικά. Θα περισσώ στα πέντε λεπτά. Βέβαια θα και ο Πετελίζη μετά να πει και αυτός από τη δική του σκοπιά Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι σημαντικό νομοθέτημα το κείμενο της Κομισιόν, αποτελεί χρήσιμη αφετηρία, αλλά νομίζω ότι θα θελήσουμε να το βελτιώσουμε. Όταν το συνέταξε το κείμενο η Κομισιόν, ίσως ορισμένα στοιχεία να μην ήταν τόσο σαφή όσο είναι σήμερα, ε, ελπίζω ότι οι τροπολογίες μου θα γίνουν δεκτές και από πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, η δομή του κειμένου δεν έχει λογική. Αυτό λέω πρώτα. Ακολουθώ τώρα τη λογική του κειμένου της Κομισιόν για να καταστεί ευκολότερο για σας να κατανοήσετε διάφορα κεφάλαια. Στο τέλος όμως θα σας εξηγήσω πώς νομίζω ότι πρέπει να διαρθρωθεί το κείμενο. Ας αρχίσουμε λοιπόν με το κεφάλαιο 2 για την επανεπεξεργασία των ε, ε, συσκευών. Έχουμε έναν ορισμό για τη μοναδική χρήση αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια επανεπεξεργασία της μοναδικής χρήσης, κάτι το οποίο είναι, ε, δεν είναι λογική. Δηλαδή, η κατάσταση εάν ορίστε κάτι ως single use, σημαίνει μιας χρήσης για έναν ασθενή σε μία θεραπεία. Ε, έχουμε και αυτό το reprocessing βεβαίως, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιπτώσεις σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, άλλες φορές υπερβάλλω λίγο, στην κουζίνα του νοσοκομείου. Έχουμε λοιπόν άλλο ορισμό μοναδικής χρήσης ή μιας χρήσης και πολλαπλών χρήσεων που είναι καλύτερο μέσα στο κείμενο. Όλα τα υπόλοιπα όσα δεν είναι μιας χρήσης θα πρέπει να είναι πολλαπλών χρήσεων. Η Κομισιόν για όσα γίνονται reprocessed προβλέπει μια διαδικασία κατασκευής για τον ε, ε, ε επανεπεξεργαστή ας πούμε έτσι αλλά πρέπει να είναι σαφές μεταξύ μας τι σημαίνει μιας χρήσεως Σημαίνει πάντα μόνο μιας χρήση. Είναι ρεαλιστικό αυτό. Όταν έχουμε ας πούμε μία κάμερα που κοστίζει 1000 ευρώ και που είναι από αυτές οι μικρές που εξετάζουν την καρδιά. Γνωρίζουμε ότι σε 90% των περιπτώσεων, ακόμα και αν θεωρείται ε, συσκευή μιας χρήσεως, θα τύχει επανεπεξεργασία. Άρα πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουμε αυτό και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει απολύτω κανένα κίνδυνο νοσοκομιακή λοιμόξεω ή άλλων παρενεργειών. Γι' αυτό παρακαλώ την Κομισιόν να υποβάλει άλλε καλύτερε ιδέε από ό,τι περιλαμβάνει στο κείμενο. Μετά, να δούμε πώ διατίθεται το προϊόν στην αγορά και τι είναι απαραίτητο. Η Κομισιόν στο κεφάλαιο 4, παράρτημα 6, λέει για τα, για τα όργανα προς τα οποία γίνεται η κοινοποίηση. Notified bodies. Θα δούμε ποια καθήκοντα θα έχουν οι οργανισμοί αυτοί, οι φορείς αυτοί. Θα εξετάσουμε και την κατάσταση από άποψη τελών. Δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των χωρών μελών ή και μέσα στις χώρες μέλη σχετικά με τα τέλη που χρεώνει ένας ε, ε, οργανισμός προς τον άλλο. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα. Κάτι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικό και πιο αυστηρό για το προσωπικό. Δεν υπάρχει σαφής υποχρέωση τώρα για οποιοδήποτε notified body και για τις τέσσερις κατηγορίες, κατηγορία 1, 2 και 3B, δεν έχουν υποχρέωση να έχουν ε, στο προσωπικό τους, φαρμακολόγους, γιατρούς κτλ. Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Πρέπει να έχουν τεχνογνωσία in-house. Όποιος θέλει να κοινοποιήσει κάποιο για το τεχνολογικό προϊόν πρέπει να έχει στην επιχείρηση ή στον οργανισμό την τεχνογνωσία, τη σχετική τεχνογνωσία. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε και τις συμβάσεις που έχουν και τις συμβάσεις που δίνουν όταν αναθέτουν για την τεχνογνωσία. Πρέπει να είναι διαφανές, πρέπει να κοινοποιείται στους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς και να διατίθεται και η επιτόπου τεχνογνωσία για να μπορεί να ελέγχει και η τεχνολογία που έρχεται έξωθεν. Για το προσωπικό και τους υπεργολάβους λοιπόν πρέπει να είναι σαφές ότι είναι εξασφαλισμένοι η τεχνογνωσία. Για το 5.1 τώρα και για το παράδειγμα 7 είναι η ταξινόμηση, classification. Έχουμε για την ώρα τέσσερις κατηγορίες. 1, 2α και 3 και 3β. Δεν με, δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα να το κρατήσουμε. Εκεί όπου διαφωνώ είναι ορισμένα άρθρα που έχει περιλάβει η Κομισιόν για την αλλαγή κατηγορίας ορισμένων προϊόντων και κυρίως τα άρθρα 19, 20 και 21. Νομίζω ότι ήδη πέρασαν τα 5 λεπτά. Α, μια τελευταία φράση. Το σύστημα έγκρισης. Ματίας πρόκειται για μεγάλο νομοθέτημα και 5 λεπτά είναι λίγο στενό κορσές. Η έγκριση λοιπόν ε, των τεχνολογικών προϊόντων για την κατηγορία του υψηλότερου κινδύνου χρειαζόμαστε conformity assessment που να είναι και μια έγκριση προ διάθεση στην αγορά, όπως είπα για την υψηλότερη κατηγορία. Οπότε δεν χρειαζόμαστε τον μηχανισμό ελέγχου γιατί η Κομισιόν στο κείμενό της δεν έχει προβλέψει pre-market authorization. Έχει όμως ένα πολύ περίπλοκο μηχανισμό ελέγχου που τον βάζει μετά. Άρα μπορεί να διαγραφεί το άρθρο 44 εάν έχουμε pre-market authorization. Και για τις κλινικές εγκρίσεις, ναι, ναι Νίκολα, τι να κάνουμε, πολύ λίγο χρόνος. Τέλος, έχω μια διαφορετική, ε, θα έλεγα στην αρχή της εγκρίσης, μετά της εγκρίσης προαγοράς, μετά επανεπεξεργασία των συσκευών μιας χρήσεως και μετά την κοινοποίηση στους οργανισμούς και τα λοιπά, τεχνογνωσία επιτόπου και να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν επαρκείς κλινικές ενδείξεις και ούτω Αυτά και λαχάνιασα. Πιο γρήγορα δεν μπορώ. Το αναγνωρίζει ο Διερμηνέας ότι πιο γρήγορα δεν θα γινόταν. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή των 5 λεπτών. Έχουμε τώρα τους και οδησίγητες. Ξέρω ότι είναι μεγάλο το θέμα, αλλά με αυτή την αναστάτωση της ημερήσιας διάταξης σήμερα έχουμε λιγότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαγκίνες, αν είναι δυνατόν, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Συμπάσχω μαζί της για το λίγο χρόνο που είχε. Είναι λίγο άδικο να ζητάει με ένα τέτοιο τεχνικό κείμενο να το συμπτύξουμε σε τόσο λίγα λεπτά. Ένα από τα βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει να ε, απαντήσετε με περισσότερο χρονικό διάστημα ε, είναι το σύστημα έγκρισης πρώτης διάθεσης στην αγορά είναι ένα σημείο κλειδί. Ακόμα δεν έχω πιστεί. Θα ήθελα να μου πείτε πώς θα λειτουργούσε ένα τέτοιο σύστημα. Δεν είμαι πεπισμένη ακόμα ότι ε, θα πρέπει να αρνηθούμε την ιδέα μιας ε, πολύ, ενός πολύ ισχυρού, ε, πολύ αυστηρού ελέγχου κατόπιν της διάθεσης στην αγορά. Νομίζω ότι εκεί έχετε απομακρυνθεί πολύ από την πρόταση κομισιών και θα ήθελα να μου εξηγήσετε γιατί και πώς θα λειτουργούσε το σύστημα. Δεύτερον, ε, για την ε, ε, ε επανεπεξεργασία και για την μία χρήση, προφανώς συμφωνώ μαζί σας, υπάρχει ένα θέμα και γλωσσολογικό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε επίσης είναι ένα τεράστιο έργο με πολύ μικρή χρηματοδότηση. Τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη προφανώς, αλλά πολλές από τις αρμόδιες αρχές δεν διαθέτουν ούτε την αρμοδιότητα, ούτε την τεχνογνωσία για να ε, κάνουν όλους αυτούς τους ελέγχους. Συνεπώς υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Ας δούμε τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς που, προς τους οποίους γίνεται κοινοποίηση, ε, γιατί είναι πολύ σημαντικά στοιχεία κλειδιά και για τη λειτουργία του τομέα και για την ασφάλεια. Συνεπώς θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτού του φορεί που ε, δέχονται τι κοινοποιήσει, Θα πρέπει να έχουν τεχνογνωσία εκεί στους τομείς ε, που ε, δίνουν πιστοποίηση και εκεί τίθεται και το εξή ερώτημα. Έχουμε στην Ευρώπη επαρκή τεχνογνωσία συνολικά και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν αυτοί οι πυρογνωμονές Ε, επίσης, είναι κανονισμός, πολύ καλό αυτό, πολύ καλή τρόπο οδηγία. Πιστεύω ότι από όλες τις πλευρές υπάρχει η επιθυμία να βελτιώσουμε το κείμενο και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει και ένα ε, χρονικό πλαίσιο 4-5 ετών πριν να αρχίσει να εφαρμόζεται το κείμενο. Ε, ξέρω ότι ξεπερνά το χρόνο μου, να σας πω όμως και δύο ακόμα πράγματα. Πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού και των ασθενών και να εξασφαλίσουμε και τη δυνατότητα της, ε, του κλάδου να καινοτομεί και να θέτει καινούργια προϊόντα στην αγορά. Θα ήθελα λοιπόν ο, η συγκήτρια να μου δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το βασικότερο θέμα που σας ανέφερα και μετά η Κομισιόν να μας πει την ε, ε, γνώμη της για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθούν τώρα Edith Estrella, Peter Liese und Anna Rosbach. Habe ich jemanden vergessen? Μήπως ε, άφησα κανέναν απ' έξω, Σνέλχαρτ. Σνέλχαρτ λοιπόν. Και για την ώρα κλείνουμε. Κράμερ. Είναι στην ουσία αδύνατο, λόγω της περιπλοκότητας του θέματος, Η Ντάγμα τα κατάφερε σε πέντε νταγμαρολεπτά, α το πω έτσι, με την ταχύτητα που είναι σε θέση να ομιλήσει. Αλλά εν τέλει καλούμαστε να αριθμίσουμε νομοθετικά προϊόντα ιατροτεχνολογικά, την έγκρισή τους και βεβαίως και τις διασυνδέσεις μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών και άλλων φορέων. Συμφωνώ με τα όσα είπε η συγγήτρια για το θέμα του ορισμού. Είμαι απόλυτα σύμφωνος. Νομίζω επίσης ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί, μάλλον να αποφευχθεί ανταγωνισμός μεταξύ των notified bodies, των ε, φορέων προς τους οποίους γίνεται η κοινοποίηση. Και νομίζω ότι όντω η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή βάση. Κάθε απόφαση κεντρικής έγκρισης. Πρέπει πρώτα να τη σκεφτούμε καλά γιατί υπάρχει η διεθνής εμπειρία στις Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει μια τέτοια συγκεντρωτική ας πούμε κεντρική έγκριση που δεν βοήθησε ωστόσο στον να αποφευθεί το πρόβλημα με τα εμφυτεύματα που προέκυψε και που είναι γνωστό το σχετικό σκάνδαλο. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί η ποιότητα των notified bodies και όλα τα notified bodies θα πρέπει να κάνουν τα πάντα ή θα πρέπει να εξειδικευθούν με ιδιαίτερες απαιτήσει, για παράδειγμα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 3 να δούμε πόσα και ποια εμφυτεύονται το στο ανθρώπινο σώμα και τι ειδικέ απαιτήσει πρέπει να ικανοποιούν όχι απλά με μια σφραγίδα ή με τα έγγραφα που παρέχει η εταιρεία, ε, ειδικά για προϊόντα της κατηγορίας 3, πρέπει να γίνουν πραγματικά, πραγματικές δοκιμασίες, real life test. Ίσως και στην Ευρώπη να χρειαστεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα, αλλά δεν επιτρέπεται τίποτα να καταλήγει στην αγορά χωρίς προηγουμένως να γίνονται δοκιμασίες υπό πραγματικές συνθήκες. Επίσης πρέπει να είναι σαφές ότι άλλο ένας επίδεσμος και άλλο ένας βηματοδότης. Πρέπει να δούμε ποιες απαιτήσει πρέπει να ικανοποιούν, ποιες είναι οι ιδιαίτερες απαιτήσει για ιδιαίτερα προϊόντα και αυτές να, είναι, να επιβάλλονται στα notified bodies. Εν τέλει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσει αυτή η pre-market authorization όπως είπε η Βρετανίδα συνάδελφός μου, χρειάζεται εποπτεία της αγοράς. Για να δούμε, υπάρχουν ενδεχομένω κάποια... Υπάρχουν κάποιες ε, παρενέργειες ενδεχομένως από προϊόντα τις οποίες δεν έχουμε διαπιστώσει πριν από τη διάθεσή του στην αγορά. Ευχαριστώ κύριε Κράμπερ. Η κυρία Άουκεν. Ο κ. Ο Σκιώδης δεν είναι εδώ και γι' αυτό, ή Σκιώδης μάλλον, και θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα εξ ονόματής της. Από όσο ξέρω, έχουμε συμφωνήσει σχεδόν σε όλα. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα στοιχεία. Ε? Ε, ο Μισελ Ριβασί έκρινε ότι μιλάμε για τρία μηχανήματα τα οποία δεν θέλω να ορίσω εκ των προτέρων. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε ορισμένα ε, σκάνδαλα και στη Δανία σε σχέση με το PIP που προαναφέρατε. Ως προς τις ε, κλινικές ε, έρευνες θέλουμε διαφάνεια ε, όχι απόρριτο, δηλαδή κανονικές διαδικασίες αδειοδότησης, έτσι ώστε να μην υπάρχει κακοδιαχείριση. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν ασφαλείς έλεγχοι και αυτό αφορά και την προσβασιμότητα στα στοιχεία, όχι μόνο στη σύνοψη έτσι ώστε να πούμε στη βιομηχανία ότι αν μπορούν να μας δώσουν μια σύνοψη, τότε μπορούν να μας δώσουν και λεπτομεριακά στοιχεία, διότι αν δεν έχουν τα στοιχεία δεν μπορούν να φτάσουν καν σε σύνοψη. Άρα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία, αν έχει γίνει σωστή εργασία ως προς τη σύνοψη του προϊόντος. Ως προς τις ε, τοξικολογικές ε, μελέτες για τα εμφυτεύματα, θα ήθελα να μιλάμε για ορμονικούς διαταράκτες περισσότερο. Δηλαδή έτσι θα πρέπει να τους κατονομάζουμε. Αυτή είναι η δική μου υπόδεξη, δηλαδή να μιλάμε για ορμονικούς διαταράκτες. έτσι ώστε να υπάρχει πραγματικός έλεγχος ως προς αυτές τις ουσίες. Ευχαριστώ. Άννα Ρόσμπαχ, η οποία αντικαθιστά την κυρία Γιανακουδάκη. Θα μιλήσω δανέζικα, μια και έχω την ευκαιρία. Μιλώ εξ ονόματος της κυρίας Γιανακουδάκη, όπως είπε και ο πρόεδρος. Η Κομισιόν πραγματικά με αυτή την πρότασή της ε, είναι πολύ επικαιρή, ε, διότι ε, πολλά σκάνδαλα έχουν πλήξει την Ευρώπη τελευταία. Και αυτό έχει οδηγήσει σε απώλεια. Έχει προκαλέσει απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού. Και απώλεια την οποία θα πρέπει να, να κτίσουμε. Η ασφάλεια του ασθενούς θα πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημα. Θα πρέπει επίσης να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να ενισχύσουμε τους ελέγχους. Επίσης θα πρέπει να ε, γίνονται ε, ευνίδιοι έλεγχοι, όχι μόνο προγραμματισμένοι. Είναι πολύ σημαντική επίσης οι κοινοποιούμενοι οργανισμοί, οι οργανισμοί οι οποίοι δέχονται τις κοινοποίησεις. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα τα προϊόντα αυτά ε, και τους κινδύνους που μπορεί να αποτελούν όπως το TUV στην Γερμανία. Ε, επίσης υπάρχουν προβλήματα με τους βηματοδότες, με τα εμφυτεύματα και με άλλου τύπου ε, προϊόντα. Είναι επίσης σημαντικό ο ασθενής να γνωρίζει όλα αυτά τα στοιχεία αυτό όμως δεν προκύπτει άμεσα από το κείμενο της Κομισιόν. Θα πρέπει στο κείμενο της Κομισιόν ε, να κάνουμε ε, ιδιαίτερη μνήμα και με αυστηρό τρόπο στα προϊόντα τα οποία επαναχρησιμοποιούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητά τους. Ιδιαίτερα αν θέλουμε να επαναχρησιμοποιούμε πολλές φορές ε, ένα τέτοιο προϊόν. Ευχαριστώ. Κύριε Στρέλα, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Dagmar για την εξαιρετική δουλειά της και για την ε, πολύ καρποφόρα συζήτηση που μας βοήθησε να κάνουμε και με τις ακρόασεις που διοργάνωσε. Ε, παρεμβαίνω ως εισηγήτρια της έκθεσης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Θα μιλήσω λοιπόν για το θέμα αυτό από την πλευρά της ασφάλειας των εργαζομένων και των χρηστών τα, ε, τα τεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως μέσα σε νοσοκομεία από επαγγελματίες του τομέα υγείας ε, αλλά και, από, ε, και μέσα σε φυλακές και άλλου τύπου περιβάλλοντα. Συνεπώς υπάρχουν κίνδυνοι όχι μόνο για τους ασθενείς αλλά και για τους εργαζόμενους τομέα υγείας που χρησιμοποιούν αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για, τους, ε, και για το βοηθητικό προσωπικό, για παράδειγμα προσωπικό ασφαλείας, ε, ε καθαρισμού, ε, στα πλυντήρια ε, κλπ. Είναι στόχοι λοιπόν και αυτής της πρότασης. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω ε, τον στόχο ποιότητας και ασφάλειας με τον ε, στόχο βελτίωσης ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Αυτός ο τελευταίος ε, στόχος επιτρέπει τη σύνδεση με την ισχύουσα νομοθεσία περί ασφάλειας στον χώρο εργασίας και έχει σχέση με το πλαίσιο αποφυγής τραυματισμών από αιχμηρά εργαλεία σε νοσοκομεία και άλλου τύπου εγκαταστάσεις. Ε, όπως βλέπετε, ο βασικός στόχος δική μου έκθεσης θα είναι να διασφαλίσουμε ότι τα ιδιωτικά προϊόντα ε, θα βελτιώσουν την ασφάλεια ε, στο χώρο εργασίας. Ευχαριστώ. Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ιδιαίτερος και την Dagmar Ροτ Μπέρεντ. Όντως το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η επιτυχία της που μπόρεσε να το αναπτύξει έστω και σε χονδρικές γραμμές μέσα σε 7 μόλις λεπτά. Εγώ κάνω τα ιατροδιαγνωστικά και βεβαίως υπάρχει διασύνδεση με το θέμα της ε, Dagmar Roth-Berendt. Πολλές από τις ιδέες τις βρίσκω χρήσιμες τις ιδέες της, να αλλάξει η σειρά των κεφαλαίων, να μπουν κάποια πράγματα στην αρχή, να βελτιωθεί η ποιότητα των ε, notified bodies κλπ. Σε αυτά συμφωνούμε. Ευχαριστώ και την κυρία Μαγκίνε, ωστόσο, σκιώδη ηγέτρια του Λαϊκού Κόμματο, που λέει ότι δεν είμαστε ακόμα απόλυτα πεπισμένοι και δεν ξέρουμε αν θα πιστούμε κιόλα ότι όντω χρειαζόμαστε pre-market authorization, δηλαδή έγκριση πρώτη διαθέσεως στην αγορά από κρατικές αρχές. Το προτείνει βέβαια μόνο για την κατηγορία 3 που είναι σχετικά περιορισμένο τομέα. Αλλά υπάρχουν και πολλά προϊόντα, υπάρχει και ιδέα μάλλον ορισμένα προϊόντα να αναταξινομηθούν από την κατηγορία 2 να πάνε στην 3 και ούτω καθεξής. Το μέγα θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει αυτό και πώς θα προχωρήσει. Θα προσθέσω κάτι σε όσα είπαν ορισμένοι συνάδελφοι. Για τα φάρμακα έχουμε την κρατική προέγκριση και πάλι τα σκάνδαλα δεν αποφεύθηκαν. Έχουμε το περίφημο φάρμακο Mediator, έχουμε και άλλα σκάνδαλα τα οποία όπως είπα δεν αποφεύθηκαν παρόλη την κρατική προέγκριση. Γι' αυτό θεωρώ ότι κατά βάση θα πρέπει να σεβαστούμε την δομή του κειμένου της Κομισιόν. Και ως εισηγητής για τα διαγνωστικά αυτό θα κάνω, αυτό θα προτείνω δηλαδή. Και για τα PIP δεν είχαμε πρόβλημα εγκρίσεως, αλλά πρόβλημα μετά την έγκριση. Εξαπατήθηκε η αρχή όπως μπορούσε να εξαπατηθεί και εξαπατήθηκε άλλωστε το notified body. Και όπως είπε και ο Κράμερ, χρειαζόμαστε, ο κύριος Κράμερ, ο Holger Κράμερ, χρειαζόμαστε real life test, δηλαδή δοκιμασίες υπό πραγματικές συνθήκες, όχι μόνο να ε, γίνεται η εξέταση επί των εγγράφων, αλλά ολόκληρη, ολόκληρη την αλυσίδα χρήσεως του προϊόντος. Αυτό είναι ένα σημαντικό το οποίο προτείνει η Κομισιόν και οφείλουμε να το ενισχύσουμε. Ευχαριστώ αγαπητέ Λίζε, η κυρία Άλντα Σούσα. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, εξαιρετική αυτή εργασία και workshop της Dagmar στις 28 του μηνός σε σχέση με αυτό το τομέα. Θα ήθελα να πω και εγώ μερικά πράγματα επί του θέματος. Καταρχήν, το θέμα της ασφάλειας των ασθενών είναι ύψης της σημασίας για εμάς και δεν νομίζω ότι είναι κάτι ασύμβατο με, τον, με την καινοτομία. Θα πρέπει όμως να υπάρχει μία νομοθεσία που να εγγυάται την ασφάλεια και όπως είπε και ο Πίτερ Λίζε, θα πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι ως προς την ασφάλεια και τους ε, όρους εφαρμογής ακόμα και μετά την αδειοδότηση κυκλοφορίας δηλαδή του προϊόντος στην αγορά. Αρκετές πτυχές της πρότασης ε, της Επιτροπής σε σχέση με την ταξινόμηση θα πρέπει να αναθεωρηθούν για να είμαστε πιο συνεπείς και θα πρέπει να υπάρξει πληροφόρηση προς το κοινό. για το τι είναι διαθέσιμο ως προς τα δηλαδή ε, ιατρικά μηχανήματα και γενικότερα να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού αλλά και όσους εργάζονται στον τομέα της υγείας. θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα για αξιολόγηση, γιατί πολλές φορές ε, πρέπει να μπορούν να προβούν και σε υποδείξεις ως προς αυτά τα medical devices. Επίσης η αναθεώρηση των δεδομένων δεν αρκεί, της περιγραφής δηλαδή των μηχανημάτων, θα πρέπει να ξέρουμε τι αποσύρθηκε, τι δεν αποσύρθηκε, τι λειτουργεί καλώς και τι όχι. Αυτά εκ πρώτης όψεως, αλλά θα έχουμε πολύ χρόνο να μπορέσουμε να επεκταθούμε. Δεν το ακούσατε ίσως όταν το ανακοίνωσα, δεν ήσασταν ακόμα παρούσα, αλλά έχουμε περίσσει το χρόνο αγορεύσεως για τον καθένα σε δύο λεπτά. Έχετε το λόγο. Ωραία, πρώτο, άμα έχει αναλάβει η Ντάγμα Ροτμπέρεν, τότε η έκθεση θα είναι καλή. Όντω η διαδικασία είναι περίπλοκη. Παρατήρηση τη Ντάγμα χωρί μικρόφωνο. Βέβαια υποστηρίζω και τον Πέτερ Λίζε που είπε ότι για ορισμένα προϊόντα το προϊόν πρέπει να εξεταστεί και εκ των υστέρων. Αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, έχω ένα άλλο θέμα. Την επαναχρησιμοποίηση ας πούμε των προϊόντων. Σε πολλές συζητήσεις που έχω κάνει έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποια αταξία. Ορισμένοι κατασκευαστές λένε «Α, το προϊόν μιας χρήσεως, παρόλο που μπορεί καταρχήν να χρησιμοποιηθεί και, και άλλες φορές, γιατί βέβαια θέλουν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους». Τα νοσοκομεία διστάζουν. Πρέπει και εδώ να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποια τάξη. Και μου φαίνεται απαραίτητο να ορίσουμε κάποιους φορείς, όχι όμως τους χρήστες, που θα πρέπει να επιτρέπουν την εκ νέου χρήση. Γιατί για τους ίδιους ε, τους φορείς που χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά βλέπω και κάποιο οικονομικό συμφέρον. Ε, α πούμε τον καθετήρα δεν θα τον χρησιμοποιήσουν ξανά Τώρα, για τα τέλη. Είχαμε και αλλού άλλη παρόμοια διατύπωση. Μετά όμως, στην εφαρμογή, καταλήξαμε σε χάος. Έχουμε διαφορετικά τέλη, λίγα χιλιόμετρα μακριά, υπό διαφορετικές συνθήκες. Ή μάλλον υπό ίδιες ή ίσες συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν ε, θα πρέπει μάλλον να εξετάσουμε ακριβώς τι προτείνει η Κομισιόν και να ξεκαθαρίσει η Κομισιόν ακριβώς ποια πράγματα εντάσσονται στα τέλη. Αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την Ντάγμαρ. Ε, Πρόκειται να είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα Βέβαια, βασικό μας νόμονα θα πρέπει να είναι η ασφάλεια. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια, να βελτιώσουμε τις προτάσεις. Είμαι υπέρ της ταξινόμησης, ε, δεδομένου ότι υπάρχουν προϊόντα ε, τα οποία ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι αξιόπιστα να εξασφαλίζουν την ε, εμπιστοσύνη του χρήστη ε, και υπάρχουν και ε, πολύ πιο σύνθετα και σημαντικά προϊόντα τα οποία είναι σημαντικά ενώ για την ζωή του ασθενούς όπως οι βηματοδότες και τα εμφυτεύματα συνεπώς υπάρχουν διαφόρων ειδών προϊόντα ίσως θα πρέπει να έχουμε και μια ακόμα κλάση για τα οποία, προϊόντα για τα οποία θα χρειαζόταν ε, και κλινικές δοκιμές. Έχουμε ένα αριθμό περιπτώσεων που μας έχουν καταγγελθεί, ε, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν ελαττωματικά ιατροτεχνικά λογικά προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να ανοιχνευθούν, δεν, ε, δεν εξασφαλίζεται η ανοιχνευσιμότητά τους και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στη διάγνωση όσο και παρενέργειες. Συνεπώς, ε, ε, οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ε, καταγράφονται και να παρακολουθούνται. Τώρα το VIP ήταν απάτη έτσι, δεν, είχε, δεν ήταν θέμα ασφάλειας, ήταν καθαρή απάτη. Αυτό είναι παρενθέση. Να πω επίσης ότι σε ό,τι φορά το λογισμικό ίσως θα χρειαζόταν να δούμε πώς πρέπει να καλύψουμε και το λογισμικό με αυτή την πρόταση. Τέλος, ό,τι αφορά την μονή πολλαπλή χρήση, ε, μία ή πολλαπλή χρήση, ε, πολλά, πολλά καλώδια, διακόπτης και λοιπά, την χάνουν, τυχαίνει ε, να θεωρούνται μονής χρήσης, ε, που αποτελούν απλώς ανταλλακτικά όμως ε, προϊόντα τα οποία είναι μόνες χρήσης. Θα πρέπει αυτό να το αποφύγουμε διότι αυτά μπορούν να αλλάξουν. Δεν είναι, υπάρχει λόγος ε, διακόπτες και καλώδια να θεωρούνται μόνες χρήσης. <clears throat> Eh, Ευχαριστώ. Μπορώ να υποστηρίξω τα περισσότερα από όσα προελέχθησαν. Είναι δύσκολη αυτή η οδηγία και τεχνική Υφή και είναι ζωτική σημασία να μπορούμε να συνεργαστούμε με εμπειρογνώμονε που έχουν πείρα σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν θέματα ασφάλεια διότι αυτό είναι ένα κομβικό σημείο που μας απασχολεί. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου την επικουρικότητα. Έχει σημασία να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, ιδιαίτερα ορισμένων πολιτισμικές, ιστορικές και ούτω καθεξής και δεν πρέπει να αλλάξουμε την καλή μεθοδολογία που κατέχουν ορισμένα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης προς την Επιτροπή, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό ισχύει και, στις, ε, και για τα μηχανήματα ερευνών in vitro, γιατί θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως προς τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα. Θα πρέπει να το δούμε με τους τεχνικούς, δηλαδή με εκείνους που διαθέτουν πύρα. Ορισμένοι από αυτούς δεν είναι σίγουροι κατά πόσο μπορούν, μπορούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Um, uh, Ευχαριστώ. Εντάχει, λέει η κυρία Τέιλορ, ως προς την ε, εποπτεία και την έγκριση πριν να τεθεί το προϊόν στην αγορά ή μετά. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ευεργετήματα ως προς την ασφάλεια και κατά πόσο θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός. Κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό λοιπόν τη στιγμή που αναθεωρούμε το, την κατάσταση προσωπικού στα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είπα έχουν μία ταξινόμηση τριών κατηγοριών και η τρίτη χρειάζεται έγκριση πριν από τη θέση ε, στην αγορά και αυτό αφορά ιδιαίτερα τα μηχανήματα αντικατάστασης γοφών. Γι' αυτό χρειάζεται και εποπτεία μετά τη θέση στην αγορά, διότι υπάρχουν, ελοχεύουν κίνδυνοι μετά από τη χρήση και θα πρέπει να δούμε τι κλινικά στοιχεία που έχουμε ως προς την χρήση των ε, μηχανημάτων από τους ασθενείς. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσωπικοί. Ευχαριστώ. Σαμπίν Λεκενιέ τιματάρχης της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Ο διευθυντής μου δυστυχώς, η κυρία Δέσποινα Σπανού, μάλλον η διευθύντρια μου, δυστυχώς κολλείεται, βρίσκεται σε διεθνές φόρουμ και δεν μπορεί να είναι παρούσα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τους τρεις στόχους της προτασός μας. Ενίσχυση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ενίσχυση στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα. Τρεις στόχοι λοιπόν που μας καθοδηγούν για την σύνταξη του εγγράφου μας. Θα απαντήσω στα διάφορα σχόλια που έγιναν. Αφενός στην κατάσταση πριν από την διάθεση στην αγορά και μετά. Και θα έλθω και στο θέμα της διαφάνειας. Ορισμένοι από εσά αναφέρθηκαν στο λεγόμενο reprocessing, στην επανεπεξεργασία, η επανακατεργασία των προϊόντων. Στο κείμενο της προτάσεως περιλάβαμε ορισμό των προϊόντων μιας χρήσεως, όπου φαίνεται να υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ των όρων όταν μιλούμε για επανεπεξεργασία προϊόντων μιας χρήσεως αυτό δηλαδή θα το αποφασίσει ο κατασκευαστής, ο οποίος διαθέτει το προϊόν του στην αγορά με πρόθεση αυτό να χρησιμοποιηθεί άπαξ μόνο. Αυτό μπορεί όντω να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μπορεί δηλαδή να προκύπτει κάποιος κίνδυνος εφόσον επαναχρησιμοποιηθεί, ή μπορεί να οφείλεται στο ότι ο κατασκευαστής δεν έχει προβεί τις απαραίτητες μελέτες για να μπορεί να δείξει πόσες φορές και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί το προϊόν. Έχουμε βάλει και ορισμό των κρίσιμων προϊόντων, δηλαδή για χειρουργικές διαιτητικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις επεμβάσεις καταρχήν αποκλείονται από την επανακατεργασία, επανεπεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση αν θέλετε. Εμείς βασιστήκαμε γι' αυτό στην γνώμη της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής περιλάβαμε την έννοια του reprocessor, αυτού που κάνει δηλαδή την επανακατεργασία, διότι αυτός εξομοιώνεται με κατασκευαστή, διότι αλλάζει τον αρχικό σκοπό του προϊόντος. Αυτός δηλαδή που προχωρεί στην επανεπεξεργασία εξομοιώνεται με κατασκευαστή και οφείλει έτσι να ε, συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις του κατασκευαστού. Τέλος, για να μπορέσουν ορισμένες χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν ειδικέ συνθήκες, περιλάβαμε ρήτρα που τους επιτρέπει να προβούν σε opt-out, δηλαδή να απαγορεύσουν την πρακτική της επανεπεξεργασίας ή την διάθεση του επανεπεξεργασμένου προϊόντος στην επικράτειά τους. Με αυτό το καθεστώς λοιπόν μεταφέρουμε στην πράξη τις επιστημονικές συμβουλές που μας παρέσχε η Επιστημονική Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο να διασφαλίζει και την δυνατότητα επανεπεξεργασίας, αλλά βέβαια με την απαραίτητη ασφάλεια. Δεύτερο, των ε, οργανισμών προς τους οποίους γίνεται η κοινοποίηση. Είναι μια δυναμία του παρόντος συστήματος και γι' αυτό ενισχύουμε τον ρόλο των οργανισμών αυτών βάζοντας ορισμένες διαφυλάξεις, δηλαδή επιβάλλουμε υποχρεώσεις στις αρχές οι οποίες καθορίζουν τους οργανισμούς αυτούς, ενισχύουμε σε ολόκληρο παράρτημα τα κριτήρια, με συγχωρείτε να ολοκληρώσετε λέει ο Πρόεδρος, για να υπάρχει ουδετερότητα, να είναι αποδειγμένη η ικανότητά τους, οι διαδικασίες, το προσωπικό τους κτλ. Υποβάλλουμε τους οργανισμούς αυτούς επίσης σε κοινού ελέγχους από εκπροσώπους της Κομισιόν και χωρών μελών άλλων χωρών μελών δηλαδή, και τέλος η εργασία των οργανισμών αυτών σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπόκειται και σε μηχανισμό ελέγχου. Σκρούτινη δηλαδή στα αγγλικά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όντως έχουμε ενισχύσει σημαντικά τον έλεγχο και τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν οι εν λόγω οργανισμοί. Μπορούμε να προχωρήσουμε και περαιτέρω, αλλά πιστεύουμε ναι, ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Η υπόσχεση της Κομισιόν ολοκληρώνει. Να έχουν λοιπόν ένα επαρκές επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά τα τέλη, στην πρότασή μας περιλαμβάνουμε άρθρο που θα χρησιμεύσει ως βάση για ένα καθεστώς. Παρακαλώ ολοκληρώστε. Όλοι προσπάθησαν να τηρήσουν τον χρόνο, ίσως και εσείς λοιπόν να μπορέσετε τώρα να ολοκληρώσετε. Ναι, λέει η εκπρόσωπη τη Κομισιόν. Ένα ακόμη, σχετικά δηλαδή με τους κανόνες ταξινομήσεω, προβλέψαμε τους κανόνες αυτούς ε, για να λάβουμε υπόψη μα την εμπειρία της εξελίξεως στο εθνικό επίπεδο. Έχουμε ένα κανόνα που αφορά τα προϊόντα τα οποία εισπνέει κανείς ή που χορηγούνται ε, δια του κόλπου ή σε άλλες περιπτώσεις, κανόνας τον οποίο έχουμε περιλάβει στο κείμενο για να αντιμετωπίσουμε θέματα δημόσιας υγείας, διότι θεωρούμε ότι τέτοια προϊόντα ενδέχεται να αποτελούν πηγή συγκεκριμένων κινδύνων. Ευχαριστώ. Να πείτε καλημέρα στην διευθύντριά σας, η οποία είναι και νέα στο πόστο της. Καλά θα είναι να εμφανίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε οι νομοθέτες, αντί να τρέχει στα διάφορα διεθνή φόρα. Καλημέρα λοιπόν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής μας η Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα από αυτά που είπαν ε, οι σκιώδεις και οι συνάδελφοι. Λέει η συγγήτρια, ο κύριος Κάβναχ αναφέρθηκε στο γεγονό ότι θα πρέπει να υπάρχει πραγματογνωμοσύνη. Με ακούτε, κύριε Κάβανοχ, δεν με ακούτε. Αναφέρομαι σε εσά και στα σχόλιά σας. οποιοδήποτε εισηγητής θα πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή πραγματογνωμοσύνη και γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο οργάνωσε ένα workshop ε, δύο εβδομάδες πριν όπου παρευρέθηκαν 180 εμπειρογνώμονες, πολλά μέλη και η δική μου πολιτική ομάδα οργάνωσε ένα workshop χτες όπου παρευρέθησαν 100 περίπου ενδιαφερόμενοι μέλη και ε, είχαμε πολλούς εμπειρογνώμονες και ε, άμεση μετάδοση από το διαδίκτυο. Άρα λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων και των ιατρών. Ως προς τα σχόλια των συναδέλφων, η Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών μίλησε για μια διαδικασία προέγκρισης για τα προϊόντα ύψης της σημασίας. Και όχι μόνο οι ενός καταναλωτών, αλλά και οι ιατροί, οι ορθοπαιδικοί, οι καρδιολόγοι και άλλες ειδικότητε ανέφεραν στην ακρόαση ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μία ε, κεντρική αντιμετώπιση, συγκεντρωτική αντιμετώπιση για την κατηγορία 3. Μιλάμε για ένα 3% της αγοράς μηχανημάτων και ένα 2% αποτελούν νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που αφορούν 500 με 600 μηχανήματα της κατηγορίας 3. Ε, Βεβαίως η Επιτροπή Δυνάμει του άρθρου 21 ε, έχει μεταφέρει ορισμένα προϊόντα στην κατηγορία 3, αλλά λυπάμαι ε, Σαμπίν, αυτό που κάνεις δεν είναι σοβαρό. Η υποψία μου είναι ότι δεν ήξερες τι έκανες, διότι μιλάμε για ε, τεχνητά ε, ότα στη, και τα βάζεις στην κατηγορία 3. Γιατί αν κάτι είναι φαρμακευτικό σκεύασμα δεν θα πρέπει να ενταχθεί στα μηχανήματα, διότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πληρούνται οι όροι και να δούμε ε, τι ισχύει όπως ε, στην ε, περίπτωση ορισμένων όπως αφορά ορισμένα προϊόντα και το pH τους γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι σε σχέση με τα καθαρτικά θα πρέπει να ξέρουμε πού τα εντάσσουμε. Υπάρχουν προϊόντα που είναι φαρμακευτικά σκευάσματα, άρα εντάσσονται σε αυτή τη γραμμή αποκλειστικά. Ο Πίτερ Λίζε πολύ σωστά είπε ότι αν λάβουμε το άρθρο 21 και εντάξουμε προϊόντα στην ε, ε, ε, κατηγορία 3 θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα λάβουμε υπόψη τα διάφορα υγρά τα οποία χρησιμοποιούμε σε περίπτωση για τα, για τα αυτιά, δηλαδή τις, τα διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω ότι μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, διότι αυτό δείχνει ότι έχουμε την, τις ίδιες πληροφορίες όλοι. Ως προς την ε, αδειοδότηση προθέσεως στην αγορά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερα μία εποπτεία μετά τη θέση στην αγορά, όπως προβλέπει η Επιτροπή υπάρχουν οι δοκιμές, ε, δοκιμές ζωής, γιατί όταν μιλάμε για τα εμφυτεύματα ποτέ δεν θα έχουμε αρκετά στοιχεία από τις κλινικές δοκιμές, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τη ζωή αυτών των μηχανημάτων στον ασθενή. Και αυτό θα πρέπει να το αποδεχτούμε σε πολλούς τομείς. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση και με κλινικά στοιχεία, αλλά ως προς τα εμφυτεύματα ε, εντός και επί του σώματος θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η διάρκεια ζωής τους. Αλλά για ορισμένα προϊόντα χρειαζόμαστε μια καλύτερη διαδικασία αδειοδότησης πρώτης θέσεως στην αγορά. Έχετε δίκιο όταν μιλάτε για εποπτεία, γιατί ορισμένα κράτη-μέλη έχουν άλλο τρόπο προσέγγισης ε, με βάση τις εθνικές αρχές και την εθνική διαδικασία αδειοδότησης για τα ε, φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως στη Γερμανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά προχωρούν αντίστροφα. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει επαναχρηματοδότηση μέσω της ΕΜΑ. Η θέση σε ισχύ αφορά τρία χρόνια, δηλαδή θα τεθεί σε ισχύ ε, με τρία χρόνια μετά από την έγκριση. Ως προς τους ε, φορείς κοινοποίησης, notified bodies, όλοι συμφωνήσατε για οποιαδήποτε κατηγορία, για οποιαδήποτε κατηγορία, θέλουμε να υπάρχει ε, ενδοπραγματογνωμοσύνη. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για κάποιο ιατρικό προϊόν χωρίς να υπάρχει ενδοπραγματογνωμοσύνη. Μπορούμε να προβούμε σε εξωτερική ανάθεση αν θέλουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και εσωτερική για να είμαστε σίγουροι για την νομιμότητα του προϊόντος. Δεν μπορούμε να έχουμε 20 ε, διαφορετικές θέσεις στους 80 φορείς ε, ενδοκινοτικός, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να έχετε αρκετές γνώμες για να μπορέσετε να εποπτεύσετε και να αναλύσετε. Συμφώνησα με τους ε, συναδέλφους ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ε, φορέων κοινοποίησης και θα πρέπει να έχουμε συστάδες ε, αριστείας, clusters of excellence, ε, δηλαδή ε, να ξέρουμε ότι στην Ολλανδία, στην ε, Λιθουανία ή αλλού υπάρχουν αυτά τα clusters of excellence. Πολλοί είπατε ότι πρόκειται για επικουρικότητα. Όχι, δεν είναι επικουρικότητα γιατί πρόκειται για προϊόντα που βρίσκονται σε ολόκληρη την κοινοτική επικράτεια. Ό,τι αποτελεί ιατρικό μηχάνημα στην τσεχική δημοκρατία είναι μηχάνημα και για τη Γερμανία και εν πάση περιπτώσει ο κατασκευαστής μπορεί να το πωλήσει οπουδήποτε. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν οι ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας παντού. Σε σχέση με την Μαργκερίτα Άουκεν, βεβαίως χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια στα κλινικά στοιχεία και περισσότερα κλινικά στοιχεία, άρα περισσότερες κλινικές δοκιμές. Εξ αρχής θα πρέπει να γίνει καταγραφή στα Μητρώα και μετά παρακολουθεί παρακολούθηση. Έτσι μπορούμε να προωθήσουμε τις κλινικές δοκιμές και να έχουμε πρόσβαση στα κλινικά στοιχεία. Χρειαζόμαστε ελέγχους και ευνηδίους ελέγχους κυρίως. Αλλά δεν υπάρχει κοινή πραγματογνωμοσύνη, αυτό δεν μας βοηθά. Πέτερ Λίζε μίλησε για την αδειοδότηση ε, πρώτης θέσεως στην αγορά. Δεν είναι πανάκια, το ξέρουν. Αλλά αναφέρθηκε και στα φαρμακευτικά σκευάσματα, όπου υπάρχουν σκάνδαλα και μετά τη διαδικασία αδειοδότησης. Εδώ πρόκειται για εθνική αδειοδότηση. Είτε πρόκειτο για ορμονικούς διαταράκτες, είτε για οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτό δεν είναι επιχείρημα για μια συγκεντρωτική προσέγγιση. Σύμφωνο με αυτά που είπε η κυρία Σόζα για ε, την δοκιμή αυτών των προϊόντων ως προς τη, ε, και τη διάρκεια ζωής που έχουν. Ως προς την επανεπεξεργασία. Είναι δύσκολο να το επιλύσουμε σωστά είναι σαν να θέλουμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Ένα προϊόν μίας χρήσης χρησιμοποιείται μία φορά και για έναν ασθενή. Αυτό εξορισμού. Αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε. Θέλουμε ε, μία χρήση για έναν ασθενή. Πιστεύουμε ότι ισχύει αυτό και θα το υπερασπιστούμε μπορούμε να πούμε ότι ισχύει για καρδιολογικές εξετάσεις που πρέπει να διενεργηθούν κάθε δύο χρόνια και στοιχίζουν χιλιάδες ευρώ. Θεωρούμε ότι αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Ό,τι και να κάνουμε δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Τότε θα κηρύξουμε παράνομα όλα τα νεσοκομεία. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Εάν όχι, θα πρέπει να δούμε πώς θα ορίσουμε τη μία και μοναδική χρήση αν ενισχύσουμε τον ορισμό της μίας χρήσης, τότε ο παρασκευαστής θα κατασκευάσει ένα πλαστικό σωλήνα, ο οποίος να μην μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και θα μπορούσε να ε, μεταποιηθεί και να ε, γίνει ε, επανεπεξεργασία. Ματίας, τέλος, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε εμείς. Εγώ θέλω να γίνεται σωστή επανεπεξεργασία καθώς και ε, πρότυπα επανεπεξεργασίας. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι αξιόπιστος και θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να μας δώσει ένα ορισμό μίας και μοναδικής χρήσης. Τι σημαίνει ότι ένα υλικό δεν μπορεί να τύχει επανεπεξεργασίας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, θέλουν να μην φέρουν ευθύνη, γι' αυτό μιλάνε για μία και μοναδική χρήση. Εγώ δεν έχω βρει την καλύτερη διατύπωση. Ευχαριστώ για τις τελευταίες σου ε, φράσεις. Ε, η κυρία Μακίνες έχει διαδικαστικό πολύ σύντομα και ζητώ συγγνώμη, να διευκρινίσει η Κομισιόν για μένα αυτά τα unannounced checks, τους ε, απρόβλεπτους ελέγχους ας πούμε. Ποιες εγγύσεις έχουμε εάν τροποποιήσουμε το νομοθέτημα και περιλάβουμε αυτή τη διάταξη ότι πραγματικά θα γίνει. Παρακαλώ η Κομισιόν. Ένα λεπτό. Απάντηση στην ερώτηση. Αλλιώς ξεφεύγουμε από το χρονικό πλαίσιο που έχουμε καθορίσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για θέμα το οποίο προέκυψε από το σκάνδαλο PIP, διότι η τρέχουσα νομοθεσία προβλέπει την, ε, δυνατότητα ο οργανισμός να κάνει ελέγχους χωρίς προειδοποίηση, αλλά στην πράξη γίνεται πάρα πολύ σπάνια. Εμείς προβλέπουμε τώρα υποχρεωτικά ελέγχους από τους ε, οργανισμούς προς οποίους γίνεται η κοινοποίηση, όπως είπα υποχρεωτικά, τακτικά στους κατασκευαστές, να ελέγχουν τους κατασκευαστές. Και, όπως είπα, θα γίνονται έλεγχοι χωρίς προειδοποίηση στις επιχειρήσεις και στη διάρκεια των οποίων ελέγχων θα λαμβάνονται δείγματα των ε, προϊόντων για να εξέταστον, για να ελεγχθούν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση. Στις 26 Φεβρουαρίου διεξήχθη σχετικό εργαστήρι. Σπάνια έζησα τέτοιο ε, καλά οργανωμένο εργαστήριο. Ευχαριστώ το Policy Department και όλους όσοι συμμετέσχουν. Βέβαια, δυστυχώ ήταν μικρή αίθουσα. Ήταν τόσο πολύ οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. Πραγματικά εντυπωσιακό. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η 3η Μαΐου, 3η Πέμπτου και στις 29 Μαΐου θα συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Προβλέπεται δε ψηφοφορία στις 10 Ιουνίου και κάποια στιγμή μετά θα οριστεί και η πορεία της προς την Ολομέλεια, η πορεία του κειμένου προς την Ολομέλεια. Έρχομαι στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, στην έκθεση δηλαδή του Πέτερ Λίζε που αφορά διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω διανύμει ένα πρώτο έγγραφο. Όποιος δεν το έχει μπορεί να το λάβει από τους ε, κλητήρες της αίθουσας. Έχω περιλάβει εδώ τα σημαντικότερα σημεία που θα συζητήσουμε στο σχέδιο εκθέσεως, το οποίο βεβαίως δεν υπάρχει ακόμη, όπως και της Dagmar Rothberend, ακόμα δουλεύουμε σκληρά για την σύνταξή του. Θα λάβουμε υπόψη τώρα, θα συζητηθούν σήμερα και θα τα περιλάβουμε και η Dagmar και εγώ στα σχέδια εκθέσεών μας. Αλλά για να υπάρχει μια πρώτη δομή σχετικά με το πώς σκέπτομαι να χειριστώ το θέμα. Το ζήτημα είναι δύσκολο και όσον αφορά τους όρους. Περί τίνος πρόκειται. Μάλιστα, in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πρόκειται για όλες τις δοκιμασίες οι οποίες γίνονται, όλα τα τεστ δηλαδή, τα οποία γίνονται εκτός του ανθρωπίνου σώματος, ας πούμε, από τη διαπίστωση του επίπεδου του σακχάρου που κάνει ο διαβητικός άνθρωπος μόνος του μέχρι, πολύ περίπλοκα βέβαια τεστ. Επειδή λοιπόν είναι πολύ τεχνικό το θέμα και ακόμη και οι όροι είναι τόσο δύσκολοι, δεν έχει εκδηλωθεί μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον για το θέμα. Στο εργαστήριο είπα ότι ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται για το μικρό αδελφάκι της μεγάλης έκθεσης για τα τεχνολογικά προϊόντα. Όμως μία ε, εμπειρογνώμων είπε «Α, όχι, δεν είναι το αδελφάκι, είναι οι γονείς της άλλης έκθεσης». Ο, ε, ε, τέλος πάντων ο γονιός της άλλης έκθεσης, γιατί αν δεν υπάρχουν in διαγνωστικά προϊόντα δεν υπάρχουν και τα άλλα. Για παράδειγμα είπαμε και τεστ για το HIV υπήρχε 10 χρόνια στην αγορά με σήμα EC πριν να το εγκρίνει η αρμόδια αρχή. Όμως εκφράστηκαν αμφιβολίες και υπήρχαν αναφορές που έλεγε ότι το τεστ αυτό δεν ε, διαπίστωνε ορισμένα είδη ιών που προκαλούν το HIV και επίσης ότι ορισμένες φορές τα αποτελέσματά του ήταν εσφαλμένα. Και τότε αποσύρθηκε. Γιατί ασχολούμαστε λοιπόν με αυτά. Διότι αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά και είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε στους πολίτες την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Η επικουρικότητα μπορεί να παίξει ένα ρόλο εκεί όπου οι χώρες μέλη για εθνικούς λόγους προβαίνουν σε αυστηρότερες έτη ρυθμίσει αλλά πάντω κατά τα άλλα πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή ρύθμιση. Για τα παράλληλα στοιχεία με την άλλη έκθεση τα είπα. Τώρα έχουμε και, θα έχουμε άλλη την έκθεση της Γκλένη Βίλμοντ και γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι στις ιατρικές εξετάσεις, τις κλινικές μάλλον εξετάσεις, επιθυμούμε να ενισχύσουμε την πρόταση τη Κομισιόν. Υπάρχει ένα κεφάλαιο και στη δική μου έκθεση και στην έκθεση τη Dagmar Ροτ Parent όπου θα πρέπει να υποβάλουμε παράλληλε τροπολογίε. Θα υπάρχουν και ιδιαίτερα θέματα. Η ταξινόμηση εδώ είναι διαφορετική. Δεν είναι κατηγορίε 1 έω 3 αλλά α έως δ. Θα πρέπει να συζητήσουμε τι κάνουμε και με τα λεγόμενα in-house test που αναπτύσσονται σε διάφορα ιατροτεχνολογικά Ινστιτούτα και δεν καταλήγουν στην αγορά και που είναι ωστόσο απαραίτητα για ορισμένε. Ε, ασθένειες ή νόσους, το ζήτημα τα, της λεγόμενης companion diagnostics, ε, δηλαδή οι ιατρο, ιατρικές εξετάσεις ειδικά κομμένες και ραμμένες για κάποιον ασθενή, επίσης οι αυτοδοκιμασίες του ασθενούς που τα εξισώνει ε, η Κομισιόν με τα τεστ που γίνονται στον ασθενή, για παράδειγμα στην νοσοκομιακή κλίνη. Άλλο είναι να το κάνει το τεστ ο γιατρός ή η ειδικευμένη νοσοκόμα και άλλο να το κάνει ο ε, οποιοδήποτε που δεν έχει την ειδική παιδεία. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν. Τώρα, το πεδίο εφαρμογής. Η Κομισιόν καλά κάνει και διατυπώνει ευρύτερα το πεδίο εφαρμογής. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Γενετικής λένε ότι δεν αρκεί αυτό. Υπάρχουν ορισμένα τεστ που κυκλοφορούν στην αγορά και που λένε ότι αν κάνεις το α ή το β θα χάσεις τότε περισσότερο βάρος ή κάποια συμπληρώματα διατροφής και ούτω καθεξής. Άλλο θέμα βεβαίως αν αυτά θεμελώνονται επιστημονικά. Ωστόσο έχουν επιρροή στην υγεία. Για παράδειγμα για ανθρώπους που είναι παχύσαρκοι ή ενδέχεται να είναι διαβητικοί έρχονται τα διάφορα τεστ και τους υπόσχονται τα πάντα και μπορεί να παραπλανήσουν κάποιον ασθενή, ο οποίος τελικά μπορεί να υποστεί σοβαρέ συνέπειες στην υγεία του. Πρέπει να μιλήσουμε και για τις προθεσμίες εφαρμογής. Η Κομισιόν προτείνει πενταετία για τα πολύ τεχνικά θέματα και ιδίω για μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, εφόσον αυτέ κληθούν να τα εφαρμόσουν, είναι σωστό. Ωστόσο, όταν έχουμε ένα τεστ HIV στην αγορά που δεν λειτουργεί, έχουμε πέντε χρόνια τότε για να λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν ορισμένα πράγματα να επιταχυνθούν. Δεν θα πρέπει να διαρκεί μια πενταετία για όλα αυτά τα προϊόντα. Τέλος, που έχω συζητήσει με τους ο συζητητή, η Κομισιόν ρυθμίζει αφενός την ποιότητα του προϊόντος και κάνει ένα σημαντικό βήμα. Ωστόσο, όλοι οι εμπειρογνώμονε με τους οποίους συνομίλησα από το Συμβούλιο τη Ευρώπη, από τον ΟΣΑ, οι διαφοροί επιστήμονε όπω ε, η εταιρεία ανθρώπινης γενετικής. Λένε καμιά φορά ότι είναι πολύ κρισιμότερο σε ποιο πλαίσιο ε, χρησιμοποιείται το προϊόν και πώς ερμηνεύονται ε, τα αποτελέσματα. Και μπαίνει και το θέμα της παροχή συμβουλών. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει εδώ και πολλά χρόνια πολύ ευαίσθητα τεστ, όπως για παράδειγμα για το DNA, να γίνονται μόνο μετά από παροχή ειδικών επιστημονικών συμβουλών, γιατί έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες. Γι' αυτό έχω αναθέσει νομική πραγματογνωμοσύνη. Το, το υπάρχει το κείμενο που προέκυψε από αυτή την πραγματογνωμοσύνη και στα γερμανικά και στα αγγλικά, μπορείτε να το βρείτε εδώ μπροστά στην αίθουσα, και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στην βάση του άρθρου 3 του Χάρη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων informed consent, δηλαδή συνένεση μετά από ενημέρωση, πρέπει να περιληφθεί κάποιο σχετικό άρθρο. Ένα τεστ, το οποίο ενδέχεται, μπορεί, ενδέχεται να έχει πολύ σημαντικέ συνέπειε, να ανατρέψει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, δεν μπορεί να γίνεται ανά πάσα στιγμή και με οποιασδήποτε συνθήκε, παρά μόνο μετά από ειδική ε, ε, επιστημονική συμβουλή. Και αυτό νομίζω πρέπει να αποτελέσει βάση και για μα εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, Πετελίζε η Σκιώδη εισηγήτρια. Παρακαλώ, δύο μόνο λεπτά. Äh, και έχω και τον Αλόης Πέτρελε και με τα ονόματα που μόλις σας ανέφερα. Α, η κυρία Τέιλο, ναι, ναι, είστε εγγεγραμμένοι. Σας είπα μάλιστα, σας αναφέρα το όνομά σας και δεύτερη. η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον Πέτερ Λίζε ότι πρέπει δηλαδή να προσπαθήσουμε σε ό,τι αφορά την βασική δομή των δύο εκθέσεων να προσπαθήσουμε να την κάνουμε όσο γίνεται πιο ε, παρόμοια. Ωστόσο, για την εφαρμογή δεν ξέρω γιατί έχουν βάλει τριετία σε μένα, πενταετία στην δική σας έκθεση. Εγώ νομίζω ότι και τα δύο πρέπει να προσαρμοστούν στα τρία χρόνια. Για θέματα για παράδειγμα των notified bodies της ιχνηλασιμότητας κλπ. Και αυτά πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ε, όμοιες οι ρυθμίσεις. Εν πάση δε περιπτώσει, τα notified bodies πρέπει να εγγυώνται την τεχνογνωσία, την πραγματογνωμοσύνη in-house. Αυτό ίσως οδηγήσει βέβαια σε κάποια, στη δημιουργία κάποιων ε, clusters, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογή, νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε αν αρκεί το περιεχόμενο του κειμένου. Αν θα συνδυαστεί κάποια ενέργεια των notified bodies με τους αρμόδιους οργανισμούς. Τώρα για την ταξινόμηση, οι τέσσερις κατηγορίες είναι καλύτερες από τις παλές λίστες που είχαν και για τα genetic testing, testing με ανησυχεί λίγο ότι ένα γενετικό τεστ ενδεχομένως να φορτωθεί μια άσχημη φήμη για παράδειγμα, για οικογένειες που ε, αντιμετωπίζουν ε, ενδεχόμενα μια γενετική ανομαλία, να είναι σαφές ότι και το παιδί ή και άλλα μέλη της οικογένειας ή και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπορούν να αποφασίσουν αν τελικά θέλουν να κάνουν παιδιά ή όχι, να μπορούν να εξετάσουν, να υποβληθούν σε τεστ για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια γενετική ε, δυσκολία, πούμε έτσι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα αυτή χωρίς να έχει οποιαδήποτε, οποιοδήποτε αρνητικό χαρακτήρα. Για τον έλεγχο δεν πρέπει να διαγραφεί ο κρατικός και για, το, για τα λεγόμενα notified bodies όπως είπα χρειάζεται να υπάρχει η σχετική τεχνογνωσία. Ρεμπέκα Τέιλορ. Δεν θα επαναλάβω πράγματα τα οποία ήδη ελέγχθησαν. Να σας πω ποιες είναι οι δικές μου ανησυχίες για ορισμένα ε, σημεία του κανονισμού αυτού. Σε ό,τι αφορά την, ε, τον έλεγχο πρώτης εμπορίας, δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν έχω στοιχεία για το πώ μπορεί να γίνει αυτό ε, για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τις ε, κλινικές ένδειξεις, καταλαβαίνω ότι χρειάζονται όχι μόνο για τα προϊόντα κατηγορίας D πρέπει να έχουμε κλινικές ε, δοκιμές για όλες τις ε, κλάσεις ε, διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στο μέλλον αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ και τους ασθενείς. Άρθρα 25 και 51 σε σχέση με την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά ε, την ε, εξαίρεση, την παρέκκληση, για μας στη δική μου χώρα ήταν πολύ χρήσιμο κάτι τέτοιο γιατί για καινούργους, παθογόνου ε, ε, παθογόνους οργανισμούς ε, βοηθάει, επιταχύνει την διαδικασία αντιμετώπισης τους όταν δεν υπάρχουν ήδη παλαιότερα διαγνωστικά τεχνολογικά προϊόντα. Ε, επίσης δεν είμαι σίγουρη για την εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα των προϊόντων της κατηγορίας D. Σε ό,τι αφορά τις ε, κινητές τεχνολογίες ε, θα πρέπει να δούμε πιο ε, σε μεγαλύτερο βάθος το θέμα. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 42 και 77 για τους ελέγχους μου έχουν εκφραστεί σημαντικές ανησυχίες για το πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία και το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι όταν πολλοί κίνδυνοι δεν αργούν μάλλον να εντοπιστούν μέχρι να εμφανιστούν οι κλινικές δοκιμές και τα αποτελέσματά τους περιμένω να διαβάσω την έκθεση Λίζε, την, ε, το προσχέδιο της έκθεσης Λίζε και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Oh, ε, Η κυρία Άουκεν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την ε, Επιτροπή για την εξαιρετική αυτή πρόταση. Αυτό είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να πούμε. Όταν ήμουν ασκιώδης για αυτό το θέμα, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο περίπλοκο είναι το όλο θέμα. Και χαίρομαι διότι το ανέλαβαν πολύ ε, υπεύθυνοι συνάδελφοι. Βρίσκεται δηλαδή σε καλά χέρια αυτή η πρόταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πέτερ Λίζε για την εξαιρετική του εργασία. Διοργανώθηκε ένα σεμινάριο, όπως γνωρίζετε, το οποίο ρίξε φως στην κατάσταση και θα ήθελα να πω ότι να εκφράσω και εγώ την ικανοποίησή μου όπως ο Πέτερ Λίζ. Οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις Καταναλωτών, όπως είπε και η κυρία Γένσεν, τόνισαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση και πρώτη στο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των ασθενών. Στόχος μας είναι να έχουμε κοινούς και βιώσιμους κανόνες και τα διαγνωστικά κέντρα να διέπονται από τις ίδιες αρχές παντού στην Ευρώπη. Στο σεμινάριο που διοργανώσαμε, αυτό το self-testing, οι αυτοδοκιμές, η αυτοδιάγνωση αναφέρθηκε. Εάν, ε, ε, Εάν χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα θα πρέπει να έχουμε και ιατρικές ε, γνώσεις δεν μιλάμε μόνο σε, για θέση σε εμπορία ορισμένων προϊόντων, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τη χρήση τους και να χορηγούνται και συμβουλές στην περίπτωση ε, αυτοδιάγνωσης. Γιατί οι αυτοδιαγνώσεις μπορεί να έχουν ολέθριες συνέπειες Αυτά τα μέσα είναι πολύ καλά ίσως για τους ασθενείς που θέλουν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της ασθενείας τους, αλλά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας. Άρα το self-testing θα πρέπει να είναι κάτι περιορισμένης εμβέλειας γιατί μπορεί να αποτελέσει ε, γενεσιουργό αιτία άλλων ασθενειών. Ο Πέτερ Λίζε ήταν πολύ ε, σαφής ως προς τις γενετικές ε, ε, δοκιμές. Τελειώνω, Πρόεδρε. Οι γενετικές δοκιμές είναι ύψης της ε, σημασίας. Συμφωνώ μαζί του και δεν μιλώ ως ε, Δανέζα, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μεγάλη διαφάνεια επί του θέματος. Λοιπόν, ο Πέτερ Λίζε καταρχήν. Θα ακολουθήσει ο κ. Κάμπερνοχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κ. Κάμπερνοχ. Γνωρίζω ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε δεν θα επαναλάβω αυτά στα οποία συμφωνούμε. Επικουρικότητα. Επικουρικότητα αναφέρθηκε επανειλημμένως. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να υιοθετούμε κοινέ αποφάσει, αλλά όταν υιοθετούμε μια τέτοια απόφαση θα πρέπει πάντοτε να προβληματιζόμαστε, να αναρωτιόμαστε αν το ευρωπαϊκό Πέδρο είναι το πιο κατάλληλο επίπεδο για υιοθέτηση τέτοιων αποφάσεων. Μήπως το εθνικό πεδίο είναι καλύτερο. Ε, ασφαλώς αυτός ο τομέας αφορά τη δημόσια υγεία και την, τα ιατροτεχνολογικά διαγνωστικά ε, προϊόντα σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Προληπτικά επίσης ε, διαγνωστικά προϊόντα είναι πολύ σημαντικά. Είναι επίσης πολύ σημαντικά τα ε, διαγνωστικά προϊόντα για χρόνιες ασθένειες, όπως ε, για παράδειγμα τους αυτούς που ασθενούν από διαβήτη. Ε, τέτοιου είδους διαγνωστικά προϊόντα μπορεί να προλάβουν ακόμα και τον καρκίνο μερικές φορές. Υπάρχει ένα θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων ε, και τα αποτελέσματα αυτών των διαγνωστικών ε, προϊόντων, τεστ, ε, πρέπει να προστατεύονται. Είναι δεδομένο, προσωπικό δεδομένο θα πρέπει να προστατεύεται. Το σε ό,τι αφορά το λογισμικό, αν το λογισμικό αποτελεί κομμάτι ενός τέτοιου προϊόντος, θα πρέπει να καλυφθεί από την νομοθεσία. Αλλά όχι να εφαρμόσουμε αυτό το κείμενο για διοικητικό software, software που, που ε, εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται στη διοίκηση. Ευχαριστώ κυρία Σόζα. Ο Πίτερ Λίζε ε, μας παρουσίασε πολύ επιτυχώς ε, το διακύβευμα Θα ήθελα να περιοριστώ στο θέμα των γενετικών διαγνωστικών διατάξεων και της άμεσης πώλησή τους στο κοινό. Ε, στο, σε μια συνάντηση βέβαια σκιωδών μπορούμε να συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, είναι αλήθεια ότι ε, μια οικογένεια που έχει μια γενετική ασθένεια είναι σημαντικό προκειμένου να κάνει τι κατάλληλε επιλογέ ζωή, να έχει στη διάθεσή τη τέτοιου είδου ε, διαγνωστικά εργαλεία. Όμως ε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόσβαση σε διαγνωστικά ε, τεστ αν δεν έχουμε κλινικά και εργαστριακά δεδομένα που να τα καθιστούν αξιόπιστα. Οπότε είτε πρόκειται για διάγνωση, είτε πρόκειται για ε, ε, προϊόντα τα οποία κάνουν κάποιο έλεγχο χωρίς την εμφάνιση συμπτωμάτων, πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων, θα πρέπει να έχουμε να υποστηρίζονται από επαρκή επιστημονικά δεδομένα, κλινικά και εργαστριακά. Η άμεση πώλησή του ε, στο κοινό μπορεί να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Θα πρέπει να το, ξανα, να το περισσότερο, να το συζητήσουμε περισσότερο, αλλά ε, δεν θα πρέπει, μάλλον θα πρέπει να αποφύγουμε αποτέλεσμα τα οποία θα είναι καταστροφικά για την υγεία των ανθρώπων. Αυτά και έχουμε, θα έχουμε στο μέλλον περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε με μεγαλύτερη άνεση. Ευχαριστώ. Hm. Εσείς κύριε Πέτρελε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το θέμα δεν αποτελεί μέρος ε, ευρύτερων πολιτικών συζητήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ίσονος σημασίας. Σημερίζομαι την άποψη εκείνων που ήδη υποστήριξαν κάτι τέτοιο. Πρόκειται για έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό εναλλακτικών διανοίγονται άλλες δυνατότητες για αυτοβοήθεια και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μία πιο αυστηρή ε, ρύθμιση Χαίρομαι διότι ο εισηγητής στο 114 ε, αναφέρεται σε μεγαλύτερη ευθύνη προστασίας της υγείας και ορίζει βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πορεία μας, την διαφάνεια, την, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος είναι από πλευράς εποπτικών αρχών και ε, παρασκευαστών να υπάρξει μεγαλύτερος ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων και σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων, διότι αν είναι λανθασμένη μπορεί να μας οδηγήσει σε ε, λάθος βήματα, σε λάθος μέτρα. Θα πρέπει να βρούμε το χρόνο για την ανείχνευση των σωστών ε, λύσεων. Όσον αφορά τις γενετικές δοκιμές, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται σωστή ερμηνεία των δοκιμών αυτών, να υπάρχει σωστή και τεχνογνωσία και πραγματογνωμοσύνη. Να γνωρίζουμε καλύτερα θέματα υγείας και να ακολουθήσουμε και το, την ηλεκτρονική μορφή παρακολούθησης της υγείας. Εκπρόσωπο της Κομισιόν που βεβαίω αναπληρώνει τη διευθύντριά τη, η οποία όπως μάθαμε δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρούσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την εισηγήτρια για τη σημασία της προτάσεως εφόσον είναι πραγματικά τόσο σημαντική η πρόληψη και η ας πούμε, προσωποποιημένη ιατρική για να ενισχύσουμε την ασφάλεια ενισχύοντας τους ελέγχους πρώτης διαθέσεως στην αγορά μέσω των notified bodies καθώς και των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων Αναφοράς που θα, θα αρχίσουν να παίζουν ρόλο μέσα στον τομέα αυτό. Έχουμε ενισχύσει επίσης την ασφάλεια και μετά την διάθεση στην αγορά με εποπτεία, ενισχυμένη μάλλον εποπτεία της αγοράς, βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ των χωρών μελών και βελτιωμένη ηχνηλασιμότητα. Όσον αφορά τα τεστ που επεξεργάζονται ε, οι οργανισμοί υγείας, θεωρήσαμε ότι για λόγους ασφαλείας θα πρέπει στο μέλλον να καλύπτονται τα τεστ αυτά με το επίπεδο απαιτήσεων που ποικίλει αναλόγως των κινδύνων που παρουσιάζουν τα εν λόγω τεστ. Σε ό,τι αφορά τα self-test έχουμε ενισχύσει τις σχετικές απαιτήσεις, κυρίως όσον αφορά τις οδηγίες που πρέπει να δίδονται και το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τα τεστ αυτά δεν θα πρέπει να μπορεί, δεν θα πρέπει να λαμβάνει την απόφαση χωρίς πρώτερη διαβούλευση με τον αρμόδιο γιατρό. Για τα γενετικά τεστ εξετάζουμε τα κείμενα του εισηγητού σε ό,τι αφορά την ενισχυμένη συνένεση που μας φαίνεται το σημαντικό θέμα και σημειώνω επίσης ότι για τα τεστ αυτά το κείμενο είναι ουδέτερο, δηλαδή αποσκοπεί στην ασφάλεια των τεστ αυτών βέβαια διοντολογικές ή ηθικές ε, ε ας πούμε πτυχές θα πρέπει να επαφιέται στις χώρες μέλη. Τα λογισμικά με ιατρικούς σκοπούς Ε, περιλαμβάνονται η διάταξη που έχει εισαχθεί ειδικά. Πρόκειται για λογισμικά, ιατρικά και όχι διοικητικά των νοσοκομείων. Και τέλος, όσον αφορά τις προθεσμίες, προβλέπουμε μακρότερη περίοδο στην πρόταση αυτή λόγω των σημαντικών αλλαγών που επιφέρει το κείμενο και λόγω επίσης του γεγονότος ότι σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των ε, τεστ ελέγχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές, ενώ με τον κανονισμό η κατάσταση θα αντιστραφεί και τα περισσότερα τεστ θα ελέγχονται από τα ε, notified bodies. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι πρέπει να παρατείνουμε την ε, προθεσμία έτσι ώστε να υπάρξει σχετική τεχνογνωσία. Ευχαριστώ πολύ. Πέτερ Λίζε θα προχωρήσει τώρα στις ε, τελικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξη. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας, γι' αυτό και είναι καλό που προχωρούμε μέσα σε επικοδομητικό πνεύμα για την παρατήρηση της ε, Dagmar Roth πρώτα. Και τέλος θα έρθω και στο θέμα των προθεσμιών που έθιξε η Κομισιόν. Κατανοώ ότι είναι δύσκολο να να συνταχθεί όλο το σύστημα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Εάν όντω είναι έτσι, και έχω και συγκεκριμένο παράδειγμα που σα ανέφερα προηγουμένω, άλλοι συνάδελφοι μπορούν να αναφέρουν άλλα παραδείγματα, ότι όντω δηλαδή αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Τότε, εφόσον σημαίνει αυτό, δεν μπορώ να προχωρήσω του χρόνου στι ευρωεκλογέ και να πω ότι α, θα φροντίσουμε ώστε σε πέντε χρόνια τα τεστ HIV που εμφανίζονται στην αγορά να είναι ασφαλή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Πρέπει να φανούμε ταχύτεροι και αποτελεσματικότεροι. Πρέπει να ταξινομούνται τα τεστ, να πηγαίνουν στα, στους ε, οργανισμούς προς τους οποίους γίνεται η κοινοποίηση. Αυτό όχι για τα τεστ HIV, διότι είναι πάντοτε υψηλού κινδύνου. Εγώ δεν είμαι και βέβαιος αν μπορούμε να συγχρονιστούμε 100% εννοώ με την πρόταση της Dagmar Roth Berend. Πάντως πρέπει για τα τεστ υψηλού κινδύνου να ε, προχωρήσουμε πολύ ταχύτερα. Συμφωνώ επίσης με τα όσα είπε η Ντάγμαρ για την τεχνογνωσία των αρμόδιων ε, φορέων. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν μπορεί να υπάρχει ειδικό γιατρός για κάθε τεστ, αλλά πρέπει να υπάρχουν γιατροί που να γνωρίζουν την ιατρική βιβλιογραφία και να μπορούν να κρίνουν εάν οι πληροφορίες που λαμβάνουν είναι ε, σωστοί. Μιλήσατε επίσης για τα ιατρικά τεστ. Δεν κατάλαβα την επιχειρηματολογία της Κομισιόν γιατί κάνουν την πρόταση που κάνουν. Τα in-house τεστ μέχρι τώρα δεν περιλαμβάνονται στην ρύθμιση. Τώρα υποτίθεται ότι θα ενταχθούν στην κατηγορία Δέλτα σαν να διατίθεται στην αγορά. Αν όμως μια πανεπιστημιακή κλινική κάνει ένα σπάνιο τεστ για μια σπάνια νόσο ή τροποποιεί κάποιο τεστ γιατί δεν λειτουργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ξέρω αν πρέπει τότε να περάσει από όλη τη διαδικασία. Δεν είμαι διόλου σίγουρος. Η κυρία Άουκεν μίλησε για το screening σε ό,τι αφορά τον, την κατεύθυνση ας πούμε είναι σωστό δηλαδή πρέπει να εγκύψουμε στα screening test που χρησιμοποιούν οι υγιείς άνθρωποι εάν μπορεί να διαγνωστεί στα νεογνά ας πούμε μια ενδεχόμενη νόσος η ασθένεια και αυτή να μπορεί να αντιμετωπιστεί ταχύτερα, νωρίτερα, βεβαίως αυτό είναι χρήσιμο. Όχι όμως να γίνεται ακρίτος. Πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποιημένη θεώρηση. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι κάθε τεστ της υγιής ανθρώπους είναι λάθος, αλλά πρέπει να κρίνουμε ποιες είναι οι κλινικές ενδείξεις. Ο Σάμπερνοχ μίλησε για την επικουρικότητα. Εγώ νομίζω ότι έχουμε ένα οξύ πρόβλημα ότι κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά τεστ τα οποία δεν λειτουργούν καλά και θα πρέπει να εξετάσουμε το κείμενο της συνθήκης εν τέλει. Η πρόταση της Κομισιόν είναι στέρεα, θεμελιωμένη στη νομική βάση του άρθρου 114 και του 168. Στο 114 λέει ότι οφείλουμε να εξασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο προστασίας στην ενιαία αγορά. Και το 168 μάλιστα περιλαμβάνει ιδιαίτερη διάταξη για τα ιατρικά προϊόντα και βεβαίως και για, και για την διάγνωση in vitro. Το ερώτημα είναι σε ποιο βάθος θα προχωρήσουμε. Και για το τελευταίο θέμα που έθιξαν ορισμένοι συνάδελφοι, τα τεστ DNA, δεν μπορεί να είναι δική μας, δικό μας καθήκον να ρυθμίσουμε την πρόσβαση των ασθενών ή των μελλοντικών γονιών ενός παιδιού σε τέτοια τεστ DNA. Δεν θα κρίνουμε εμείς αν θα το επιτρέψουμε ή όχι. Δεν είναι δική μας δυνατότητα αυτή. Συμφωνώ εδώ με την Τάγμαρ. Μία μικρή εξαίρεση, όπω έχει ήδη περιλάβει σε απόφασή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα γενετικά τεστ για την επιλογή φύλου του παιδιού, εφόσον δεν έχει καμία σχέση με ενδεχόμενη γενετική ανομαλία, παρά μόνο για την επιλογή του φύλου. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ίδιο το Διεθνέ Δίκαιο, άλλωστε, και οι αποφάσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη λένε τα ίδια πράγματα. Ωστόσο, καθήκον των γονιών είναι να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τη σχετική προφορία. Τώρα, προφορία να διαθέτουν. Ναι, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, μπορεί να έχει σημαντικότατες επιπτώσεις. Η κυρία Τσούσα που ασχολείται εδώ και μια εικοσαετία με την γενετική των ανθρώπων υπάρχει ένα σύνδρομο του Κορέα Χάντιγκτον το οποίο οδηγεί στην, στον θάνατο και ξεσπάει γύρω στο 50 έτος. Εάν ωστόσο το ανακοινώσω αυτό σε έναν 18χρονο, αυτό μπορεί να έχει τη. βαρύτατες συνέπειες και για την οικογένεια, του οικείου του, για την ασφάλιση. Αυτά πρέπει να τα σκεφτεί κανείς πάρα πολύ προσεκτικά για το αν θέλει καν να διαθέτει την πληροφορία αυτή. Υπάρχει και το δικαίωμα της μη γνώση, το οποίο και αυτό είναι άξιο προστασίας. Γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντικό, όπως και όλοι οι εμπειρογνώμονε, ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται σε ένα ιατρικό περιβάλλον με σωστή ε, παροχή συμβουλών, γιατί υπάρχει το πρόβλημα και ο κίνδυνος να λάβει κανείς τη γενετική πληροφορία από τρίτους για παράδειγμα από τον σύντροφο, από τον γείτονα. Αυτά τα πράγματα πραγματικά είναι αδιανόητα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν πολύ ξεκάθαροι κανόνες και σε ό,τι αφορά την χρήση των τεστ. Είναι ίσως χρήσιμο να υπάρξει ένα πλαίσιο όπου οι χώρες μέλη να μπορούν να αποφασίσουν. Αλλά το άρθρο 3, όπως είπα, προβλέπει την συνένεση μετά από ενημέρωση informed consent. Και αυτό πρέπει να διατυπωθεί μέσα σε μια ε, διάταξη ειδική και βασισμένη, όπως είπα, στο άρθρο 3. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε τη συζήτηση των θεμάτων 4 και 5. Οι τροπολογίες για την έκθεση του Πίτερ Λίζε μπορούν να κατατεθούν μέχρι το μεσημέρι της 3ης Πέμπτου. Ε, στις 29 Πέμπτου θα συζητήσουμε στην Επιτροπή μας και η συζήτηση προβλέπεται για την 17η. Το δε, η δε πορεία προς την Ολομέλεια ακόμη δεν έχει καθοριστεί. Σας ευχαριστώ και προχωρούμε στην έκθεση του κυρίου Φράνκο, Γενικό Ενωσιακό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον έως το 2020 με τίτλο «Ευημερία μέσα στα όρια του πλανήτη μας». Θα δώσω αμέσως το λόγο στον συνάδελφο και παρακαλώ να φροντίσετε όσοι δεν επιθυμείτε πλέον να συμμετάσχετε στη συζήτηση να αποχωρήσετε ησύχως από την αίθουσα ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να τα πει μέσα σε κάπως ευπρεπές περιβάλλον. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και το ρολόι. Όσοι θέλουν να λάβουν το λόγο ας τον ζητήσουν ευθύ αμέσως να σημειώσουμε τα ονόματα και θα σας ανακοινώσω τα ονόματα που θα έχω εγγεγραμμένα στον κατάλογο αμέσως μόλις ολοκληρώσει την παρουσίασή του ο κύριος Φράνκο. Πέντε λεπτά κύριε Φράνκο. Euh, Πρόεδρε, έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 26 Φεβρουαρίου για αυτό το θέμα. Ε, μετά Έστειλα την έκθεση μεταφρασμένα μάλιστα σε όλες τις ε, γλώσσες την ε, Δευτέρα. Πριν ακούσω τους ε, συναδέλφους να δούμε λίγο τις τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά το στόχο 1, προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να, προσθέσω, να προσθέσω τον όρο αξιοποίηση γιατί θα πρέπει να επιμείνουμε στην αξία αυτού του κεφαλαίου, την, να επιμείνουμε στην ανάγκη να ε, την, το αξιολογήσουμε και ενδεχομένως ε, να πληρώνουμε και αυτές τις υπηρεσίες, περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Ε, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η φύση θα πρέπει να έχει η, οικονομικό, να, η οικονομική ανταπόδοση, αλλά ο γεωργικός τομέας είναι πολύ σημαντικό να παίξει ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Είναι σημαντικό ε, να ε, ε, μην υπερνομοθετούμε, αλλά η οικολογική αιρεσιμότητα είναι σημαντική και θα πρέπει να εφαρμόζεται υπό την προπόθεση ότι η αντίστοιχη οδηγία θα εφαρμοστεί με τρόπο ισοδύναμο σε όλα τα κράτη-μέλη για να μην επιβάλλουν υπερβολικά βάρη στους ορισμένους γεωργούς. Επίσης, υπογραμμίζουμε για αυτό το στόχο την σημασία της βιοποίησης ποικιλότητα στη θάλασσα, την καταπολέμηση της μόλυνσης των θαλασσών και ε, την βιώσιμη δάσωση. Σε ό,τι αφορά ε, το έδαφος, είναι γνωστή η οικονομική κατάσταση των κρατών μελών, συνεπώς υποστηρίζω μια ρεαλιστική λύση. Ο ορισμός της εθνικής, Εθνική εθνικής στρατηγικής να ε, έχει σχέση με την μεθοδολογία ε, εντοπισμού των μεγαλύτερων κινδύνων. Ε, επιμένω επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί η επικοινωνιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά το περιβάλλον να ενισχυθεί η εκπαίδευση στην προστασία του περιβάλλοντος και να στηριχθούν οι δράσεις των πολιτών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών. Για το στόχο 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει αποτελεσματική οικονομία στην χρησιμοποίηση των ε, πόρων ανταπογωνιστική και χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Συνέργειε λοιπόν εδώ χρειάζονται ανάμεσα στη βιομηχανία, το περιβάλλον και την οικονομία. Πράσινη ανάπτυξη δηλαδή. Έχω χρησιμοποιήσει επίση την έκφραση οικολογικό New Deal στην αιτιολογική μου έκθεση. Προσπάθησα να αποδείξω την ε, σημασία η περιβαλλοντική πολιτική να γίνει μοχλός υπέρ της ανταγωνιστικότητας και υπέρ της αναθέρμανσης ευρωπαϊκής οικονομίας. Ιδιαίτερη σημασία δίδω στην βελτίωση της ε, περιβαλλοντικής επίδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την αρχή 9 της Small Business Act. Ε, και στην κατάρτιση ε, σε θέματα πράσινης οικονομίας. Ε, εισάγω και μια στοιχεία σε ό,τι αφορά την βιώσιμη κατανάλωση, την καταπολέμηση της πατάλης τροφίμων, την γενίκευση της ε, περιβαλλοντικής ε, σήμανσης των προϊόντων της ε, ε, αξιολόγησης ε, του, των επιπτώσεων της ευρωπαϊκής κατανάλωσης σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Η προθεσμία επίσης του 2020 δεν είναι ρεαλιστική, δεδομένη στις ετερογένειες των κρατών μελών. Σε επιπλέον, υπάρχουν συγχύσεις σε ό,τι αφορά το τι σημαίνουν τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε. Δεν χρησιμοποιούμε την ίδια γλώσσα στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα. Ε, ορισμένοι χώρες ε, λένε ότι ε, τα, ε, τα τα απορρίμματα, των, ε, τα οικιακά απορρίμματα δεν θα πρέπει να θεωρούνται βιομηχανικά, αλλά πολλές φορές ε, στην πραγματικότητα καταλήγουν να είναι βιομηχανικά ε, απορρίμματα. Ε, ε, η ιεραρχία προβλέπει μάλιστα και εξαιρέσεις ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων. Κατά την άποψή μου μια σημαντική πρόταση θα μπορούσε να επιτευχθεί αν τα ε, αν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και αυτά που μπορούν να κομποστοποιηθούν ε, να ε, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την προστασία α, για την, της υγείας από περιβαλλοντικούς παράγοντες κάνω ε, προσθήκες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού αέρα. Ε, η, ε, επίσης αναφέρομαι στην συνέχεια της ε, λειτουργίας του, της του REACH. Ε, επίσης, θα πρέπει να εφαρμόσουμε ε, την αρχή της εφιούς νομοθεσίας, της απλοποίησης της νομοθεσίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα περιβάλλοντος. Οι κανόνες θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται καλύτερα για να αποφεύγουμε την καταστατήγησή τους. Επίσης θέλω οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν περισσότερο γιατί αυτό θα βελτίωνε την εφαρμογή της νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά τις ε, επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, ε, ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη ε, να μετρήσουν ποιες είναι οι ικανότητές τους και να τις χρησιμοποιήσουν πλήρως. μια κοινοτική βοήθεια θα μπορούσε να ε, χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Σε σοβαρές περιπτώσεις και ε, λαμβανόμενο υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών θα πρέπει το θέμα να συζητηθεί πέραν της ε, έκθεσης αυτής. Σε ό,τι αφορά το στόχο 5, υπογραμμίζω την σημασία να βελτιώσουμε και να, ε, τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή και τις Εθνικές Αρχές Περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει περισσότερο ε, στην ε, διακυβερνητική πλατφόρμα βιοποικιλότητας. Σε ό,τι αφορά το στόχο 6, υπογραμμίζω διάφορα σημεία. Για παράδειγμα, θα, η, η χρηματοδότηση του Natura 2000, τα διορθωτικά, οι αυτοδιορθωτικές δράσεις, θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα, πρέπει να ορίσουμε καλύτερα ποιες ε, είναι οι ε, ε, επιδοτήσεις που βλάπτουν το περιβάλλον, να δούμε καλύτερα το θέμα των περιβαλλοντικών επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά το, δε, το στόχο 7, δεν έχω κάνει καμία πρόταση τροπολογίας. Για τον στόχο 8 έχω προτείνει διάφορες προσθήκες για να εντάξουμε την ε, αστική βιοπικιλότητα, την διαχείριση ενέργειας, ε, την καινοτομία την, και τις βιώσιμες κατασκευές. Σε ό,τι αφορά τον τελευταίο στόχο, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιφερειακό επίπεδο, Νομίζω ότι ε, θα πρέπει το βάρος να μοιραστεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τρίτες χώρες. Ο περιβαλλοντικός παράγοντας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Επιμένω λοιπόν στην ανάγκη αμοιβαιότητα και στην ανάγκη να καταπολεμήσουμε το περιβαλλοντικό dumping. Ως συμπέρασμα δεν ήταν εύκολο να περιορίσουμε τον αριθμό των τροπολογιών όπως γνωρίζετε. Θα ζητήσω και από τους συναδέλφους να είναι λογικοί έτσι ώστε το κείμενο αυτό να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατό. ich weiß, dass es sehr schwer ist, so Äh, Ευχαριστώ κύριε Φράνκο. Είναι πράγματι δύσκολο να ε, παρουσιάσει κανείς ένα τόσο περίπλοκο θέμα σε τόσο σύντομο χρόνο. Επίσης, αυτά είναι τα ονόματα που είναι γεγραμμένα. Επίσης και Χίπνερ. Ωραία, λοιπόν. Αυτό είναι ο καταλόγο των εγγεγραμμένων. Ο καθένα δύο λεπτά. Γιο Ο κύριο Φράνκο φάνηκε επιμελής. 75 τροπολογίε, Αγαπά τα δάση και η προστασία των δασών διαπνέει ολόκληρη την εκθεσή του. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πολλές από τις τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο της Κομισιόν βιοπικιλότητα, αστικό περιβάλλον, βιώσιμη κατανάλωση και βιώσιμη παραγωγή είναι πράγματα τα οποία υποστηρίζουμε και εμείς. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου μπορούμε να βελτιωθούμε και εκεί θα, θα κατατεθούν τροπολογίες για τα απορρίμματα. Πρέπει να τηρήσει κανείς την ιεραρχία, δηλαδή αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων, επανεπεξεργασία και εν τέλει απόρριψη. Για το έδαφος λέγονται λίγα πράγματα, νομίζω είναι κάπως αδύναμα, χρειάζεται, χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και όχι μόνο εθνικές στρατηγικές. Για το κλίμα χρειάζεται επιγόντως ενίσχυση μέσα στα πλαίσια του κόνσεπτ αυτού. Το πακέτο κλίματος 2020 πρέπει να συζητήσουμε. Η προσαρμογή, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και όλα αυτά είναι ανοιχτές πληγές για την αποδοτική χρήση των πόρων να ενισχυθούν οι στόχοι και οι δείκτες για τις επιθεωρήσεις. Κύριε Φράνκο, οι εθνικές αρχές βεβαίως οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αλλά χρειαζόμαστε και ένα κοινοτικό μια κοινοτική προσέγγιση. Η ΙΜΠΕΛ είναι βέβαια ένα όργανο που λειτουργεί όπως λειτουργεί, αλλά έχουμε και ένα σχετικό εργαστήριο την επόμενη εβδομάδα. Για τα θέματα αυτά θα καταθέσουμε ορισμένες τροπολογίες. Εν τέλει όμως σας ευχαριστώ για την καλή δουλειά που κάνατε με τις τροπολογίες σας ως εισηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γιο. Ο κύριος Χερμπράντι. Θαυμάσια δύο λεπτά για να μιλήσω για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας μας έτσι ώστε η οικονομία μας να γίνει ακόμα πιο βιώσιμη και αυτό αφορά και το ε, έβδομο περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να φέρει τον τίτλο περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόγραμμα. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε πιο αποδοτικοί με τους πόρους που διαθέτουμε στον πλανήτη μας, ε, αυτό θα αποτελέσει ε, ένα μεγάλο μέρος του, του γενικότερου στοιχείου ανταγωνιστικότητας. Ευχαριστώ τον Γκαστόν Φράγκο, συμφωνώ με πολλές τροπολογίες του, αλλά σε μερικές είμαι επικριτικός. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή δεν θα πρέπει όμως να αποκλείσουμε νέα νομοθετικά βήματα. Είναι αναπόφευκτα. Προτεραιότητα υπαριθμών 1, προστασία, διατήρηση και προώθηση του φυσικού μας κεφαλαίου. Εδώ μιλάμε για τη γη και τον υδάτινο ορίζοντα, τον υδροφόρο ορίζοντα. Γι' αυτό ε, δεν δέχομαι τις τροπολογίες που αποδυναμώνουν κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι η οδηγία πλαίσιο θα πρέπει να μας διέπει. Ο δεύτερος στόχος αφορά την οικονομική πτυχή του θέματος. Ο εισηγητής διαγράφει την απόλυτη αποσύνδεση ε, χρήσης και χρησιμοποιεί το κριτήριο του ΑΕΠ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Υπάρχουν ε, βεβαίως ε, διαφορές μεταξύ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά ορισμένες επικεφαλής χώρες ε, δεν μπορούν να προχωρήσουν ε, γιατί δεν υπάρχει μια ευφυής διαχείριση στις χώρες που μένουν πίσω. Τέλος, επειδή έληξαν τα δύο μου λεπτά, η προτεραιότητα υπαριθμών 6 για τις επενδύσεις στην πολιτική περιβάλλοντος και υπέρ του κλίματος Νομίζω ότι ε, εδώ ε, πρόκειται για έναν απαράβατο όρο. Ας ε, χρησιμοποιήσουμε τον όρο του ΩΣΑ και ας αρχίσουμε να ας ασχοληθούμε με την βαθμιαία απόρριψη αυτών των επιδοτήσεων. Η Μαργαρίτα Άουγκεν είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ ε, δεν είναι ότι πιο αυτονόητο μέσα σε δύο λεπτά να καλύψω το ευρύ αυτό θέμα. Καταρχήν ευχαριστώ τον Γκαστόν Φράνκο, τον εισηγητή και όταν πρέπει να βρούμε συμβιβασμούς, προτάσεις συμβιβασμού είναι μία μπορώ να πω ευχάριστη διαδικασία. δεν θα πρέπει να μιλάμε για κατασπατάληση ε, πόρων. Θα πρέπει πάντως να γίνεται ε, καύση αποβλήτων τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρξει άλλος τρόπος απομάκρυνσης. Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί. Δεν ε, είναι αυτονόητο στην Επιτροπή Αναφόρων Έχουμε πολλές προσφυγές πολιτών, πολλές αναφορές. Ελπίζω, Γκαστόν, να καταλάβεις ότι χρειαζόμαστε και την υποστήριξη των πολιτών. Βεβαίως, η Επιτροπή επίσης θα πρέπει να ε, δράσει στο επίπεδο, σε επίπεδο περιβάλλοντος. και πιστεύω ότι η σύμβαση του άρχους θα πρέπει να ισχύσει πλήρως, δηλαδή να μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και οι πολίτες. Αυτό είναι προαπαιτούμενο. Μιλώ για προοδευτικά βήματα αντιμετώπισης των θεμάτων. Μιλάμε για το Business Europe και για το Business Europe Act και ε, δεν θα πρέπει να καταρακώσουμε αυτή την καινοτόμο ε, βιομηχανία. Ελπίζω, Γκαστόν, να τα καταφέρεις να γίνει αυτό ευρέως κατανοητό, ότι θα πρέπει να έχουμε με το μέρος μας ε, τις καινοτόμες βιομηχανίες και στον ε, κλιματολογικό τομέα θα πρέπει να τα καταφέρουμε. Ja, ja, Νομίζω ότι και εδώ πρέπει να καλύψουμε τόσα θέματα, κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Ευχαριστώ τον Γκαστόν Φράνκο γιατί εργάστηκε επί μακρόν επί του σχεδίου. Ε, βεβαίως, ε, αρχικά το κείμενο ήταν διαθέσιμο μόνο στα γαλλικά, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση ε, μεταξύ στόχων και μέσων. Ελπίζω να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ε, ενδεχόμενη επίτευξη των ε, στόχων. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους αλλά και κριτήρια για να αποτιμήσουμε το μέλλον. Το έβδομο πρόγραμμα δράσης ε, θέλει να περιορίσει τους εμπλεκόμενους τομείς θα πρέπει να επικεντρώσουμε την ε, προσπάθειά μας σε συγκεκριμένους τομείς, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης. Ο κύριος Φράνκο μίλησε για τον θαλάσσιο τομέα, το τομέα των θαλάσσιων πόρων και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για τη διατροφική ε, αλυσίδα δεν θα πρέπει να γίνεται καύση των ε, τροφικών αποβλήτων. Θα πρέπει να γίνεται μεταποίησή τους κατά κάποιο τρόπο. Η ανακύκλωσή τους, ανακύκλωση αυτών. Ε, ίσως θα πρέπει να το συνδυάσουμε αυτό με άλλες οδηγίες, δηλαδή πόντιση, διάθεση, ε, δέσμευση, απομάκρυνση. Ως προς τη διεθνή πτυχή του θέματος, οι και τρίτες χώρες και οι χώρες του τρίτου κόσμου θα πρέπει να συνδράμουν, γιατί χρειαζόμαστε οι μεν τους δε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Δύο λεπτά έχετε κυρία μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα οι πολίτες μας κοιτούν το νέο πολιετές πρόγραμμα πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αναρωτιόνται πόσα χρήματα θα διατεθούν για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τη δουλειά του οι συνάδελφοι μίλησαν για την επεξεργασία των απορριμμάτων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα διότι δεν λύνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται ασφαλώς να εκπαιδευτεί το κοινό και να καταλάβει την σημασία της περιβαλλοντικής πολιτικής έτσι ώστε να συμμετάσχει ενεργά. Θα πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα στους πολίτες μας. Στην αιτιολογική εκθεσή αναφέρεται πως ο μεγαλύτερος αριθμός παραβιάσεων της ευρωπαϊκή Νομοθεσίας εντοπίζεται στον περιβαλλοντικό τομέα. Εδώ συζητούμε για το θέμα αυτό κατά καιρού. Είναι πολύ σημαντικό η νομοθεσία που υπάρχει να εφαρμόζεται. Όχι πως δεν υπάρχουν και ένα στην νομοθεσία, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον η νομοθεσία που έχουμε να εφαρμόζεται. Και βέβαια θα πρέπει να αποφύγουμε ιστερίες, ε, όπως για Παραδείγματο, σε ορισμένε χώρε ε, μπλοκάρονται προγράμματα κάθε φορά που κάποιοι πολίτε αρχίζουν και διαμαρτύρονται. Ε, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ και οι αποφάσει που λαμβάνονται να είναι ε, ισορροπημένε. Ευχαριστώ. Yeah, Ευχαριστώ. Γκαστόν Φράγκο, δεν προλαβαίνω να σα δώσω καν συγχαρητήρια. Καλή έκθεση όμω, πραγματικά θέτεται των δάχτυλων επί των τύπων των ύλων πραγματικά χρειάζονται αποφάσεις για τον ορισμό των απορριμμάτων είναι απαραίτητος καλύτερη επικοινωνία για την διάδοση καλών θεωτικών εξελίξεων. Υπάρχουν και καλά παραδείγματα λοιπόν και αυτό το λέτε μέσα. Πολύ μου αρέσει η τροπολογία στις υπαριθμών 73 που αναφέρεστε σε μεγαλύτερη διασύνδεση με την εξωτερική πολιτική και πολιτική εμπορίου όπου ήδη έχουμε κάποιες προδιαγραφές, εκεί να περιληφθούν οι δικές μας προδιαγραφές εντονότερα. Για την προστασία του εδάφους, λέτε ότι είναι καλύτερο να ρυθμιστεί εθνικά. Εγώ θεωρώ ότι σωστό είναι αυτό, αλλά πρέπει να αναφερθούμε και στην σφράγιση του εδάφου αν μπορεί να το πει κανεί έτσι, ε, στα ελληνικά. Πάει να πει δηλαδή εκεί όπου το έδαφος κλείνεται με κατασκευή δρόμων κλπ. Και, και δεν μπορεί ούτε να απορροφήσει ύδατα τίποτε. Τώρα, αυτά τα πράγματα πρέπει να οριστούν και καλύτερα. Να είναι σαφές, εφόσον για παράδειγμα επιβάλλει κανείς κυρώσεις, να είναι μετρήσιμες. Πολλά από τα προβλήματα των νερών δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του ενός ή του άλλου. Και γι' αυτό χρειάζεται μια πιο ευαισθητοποιημένη αξιολόγηση. Εν τέλει, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εξετάζουμε τακτικά και την εφαρμογή του υφιστάμενου δικαίου. Υπάρχουν πολλοί νόμοι, πολλά νομοθετήματα που συχνά δεν ελέγχεται η εφαρμογή τους. Αυτό για μένα είναι μέγα θέμα. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την ε, εξαιρετική έκθεση. Φλόρεντς. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Γνωρίζετε τις ανησυχίες μου για αυτά τα προγράμματα δράσεων. Τα έχω ξαναπεί. Καλό μου φαίνεται ότι δεν έχετε βάλει τόσο συγκεκριμένους στόχους με συγκεκριμένα νούμερα. Γιατί αυτό, κάτι τέτοιο, πρέπει να γίνει σε επιμέρους εκθέσεις και όχι σε αυτό το πρόγραμμα δράσεων για το περιβάλλον. Νομίζω δεν χρειάζεται να βάλει κανεί νέου ποσοτικούς στόχου Για τα θέματα του εδάφους τα εξήγησε η Κρίστα Κλά και συμφωνώ μαζί της. Προστασία του περιβάλλοντος και οικονομική πολιτική πρέπει να συνδυαστούν καλύτερα. Αυτό το έχουν κατανοήσει πολλοί. Το λεγόμενο στα αγγλικά food waste, δηλαδή απορρίμματα τροφίμων. Αυτά είναι στην ουσία προϊόν για τα απορρίμματα γενικότερα. Μπορεί κανείς να συζητήσει και να διαφωνήσει για την ιεραρχία των απορριμμάτων. Βεβαίω αυτή δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Πρέπει να την σκεφτούμε από την αρχή. Όπως είναι το κείμενο της Κομισιόν, είναι λευκή επιταγή για την καύση Αυτά ίσως ήταν καλά πριν από 20 χρόνια. Έχουμε καλή καύση, αλλά δεν έχουμε καλή τεχνολογία για την ανακύκλωση. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να προχωρήσουμε σε περισσότερη σωστή ανακύκλωση και χρήση και διάθεση των υλικών που προκύπτουν από την ανακύκλωση. Η καύση δεν πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή. Βεβαίω, στο τέλο, αν δεν μπορεί να κάνει κανεί το συγκεκριμένο απόρριμα τίποτε άλλο, θα το καύσει. Πάντω λυπούμε που η Κομισιόν δεν καταφέρει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βγει και να πει ότι χρειαζόμαστε μια οδηγία για τις χωματερές. Οι Ελβετοί τα καταφέρανε καλά, πολύ καλύτερα αυτά. Βέβαια, αυτά έχουν και τυριά με τρύπε. Παρόλες τις, ε, τους δισταγμούς ε, και τις δυσκολίες, ε, κάθε μερικά χρόνια έχουμε ένα καινούριο πρόγραμμα πλαίσιο και τα θέματα τα οποία καλύπτονται προφανώς δεν σταματούν στο 2020 αλλά φτάνουν μέχρι το 2050. Έχω τα εξή σχόλια. Καταρχήν υπάρχει η εθνική νομοθεσία, το εθνικό δίκαιο, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεύτερον, πρέπει να, να δούμε καλύτερα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. οι εθνικές νομοθεσίες προβλέπουν, ε, ε, περιέχουν διάφορες ε, διατάξεις, διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε από το τοπικό μας πεδίο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται η βιομηχανία θα πρέπει να συνδέεται με την ε, έρευνα έτσι ώστε να επιλέγουμε κάθε φορά τις ε, καλύτερες τεχνολογίες και τις καλύτερες μεθόδους επεξεργασίας. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η ε, πρόθεση καινοτόμων πρωτοβουλειών θα μπορούσε να μας ε, δώσει λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων σε όλες τις ε, χώρες, όχι μόνο σε μία ή δύο. Ένας κατάλογος ε, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ. Η κυρία Χίπνερ ολοκλήρωσε τον κατάλογο των αγορητών. Για την προστασία του εδάφους, τροπολογία 16 κύριε Φράνκο, πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό. Εσείς μιλήσατε και για το ορίο συν 20, για την χρήση και για κατάχρηση των εδαφών. Εδώ όμως αποδυναμώνεται αυτό, διότι προβλέπεται στρατηγικές και όχι και όχι σε ρυθμίσεις συγκεκριμένες. Από το 2005 που είμαι ευρωβουλευτής έχω δει όλες τις λεγόμενες στρατηγικές να αποτυγχάνουν και αυτό έχει κάποια σχέση και με το επόμενο θέμα για την αυτοκινητοβιομηχανία. Χρειαζόμαστε νομικά δεσμευτική διατύπωση για να μπορεί να επιτύχει. Βεβαίως το θέμα είναι αμφιλεγόμενο και εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό κατ' επανάληψη. λιγότεροι στόχοι ε, καμιά φορά είναι καλύτερα εφόσον αυτοί οι λιγότεροι στόχοι είναι νομικά δεσμευτικοί. Αρκούμε σε αυτά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην Κομισιόν, στην κυρία Σούμαχερ που είναι επικεφαλής μονάδος στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ορίστε. Ευχαριστώ. Υποθέτω ότι ισχύει και για μένα το όριο των δύο λεπτών. Α, μπορείτε να μιλήσετε πέντε λεπτά. Δεν θα μιλήσω λοιπόν τόσο γρήγορα. Καλά. Θα συγχαρώ πρώτα τον κύριο Φράνκο για την έκθεσή του. Εκτιμούμε πολλά από τα σχόλιά του και ιδίως την προσπάθειά του να τονίσει πώς η πολιτική περιβάλλοντος βελτιώνει και την απασχόληση, ε, προστασία του, των πολιτών και ούτω καθεξής. Βεβαίως και τα θέματα της βιοποικιλότητας είναι πολύ σημαντικά και υποστηρίζουμε ορισμένες, όχι όμως όλες, από τις τροπολογίες του για τα δάση, διότι χρειάζεται κάποια ισορροπία στα οικοσυστήματα και να μην βάλουμε στο πρόγραμμα και υπερβολικά πολλά δάση. Πάντως, δεχόμαστε και πολλά από τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών, με τα οποία συμφωνούμε. Ορισμένες τώρα ειδικότερες ανησυχίες. Παρακολούθησα προσεκτικά τα όσα εξήγησε ο κ. Φράνκο για το πρασίνισμα της κοινή αγροτικής πολιτικής και το δυναμικό της κοινή αγροτικής πολιτικής. Συμφωνούμε. Άκουσα λίγο ε, στα λόγια του μεγαλύτερη ευκαμψία από αυτή που δείχνουν οι τροπολογίες του. Εμείς προτιμούμε αυτές τις διατυπώσεις, τουλάχιστον εφόσον προέρχονται από τη δική σας Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό είναι σημαντικό για το πρόγραμμα. Οι κύριοι Λάινεν και Γκρότε με καθησύχασαν για το θέμα του εδάφους. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε όλα όσα λέει ο εισηγητής στην 16, στην του 16. Χρειαζόμαστε νομική δεσμευτικότητα βέβαια. Υπάρχει και το στοιχείο αυτό για να επιτευχθούν και οι στόχοι τη βιοποικιλότητας κλπ. Διότι χωρί δεσμευτικό, όπω εξηγήσατε και εσεί, περιβάλλον δεν πρόκειται να ε, επιτύχουμε. Συμφωνούμε και εμεί σε, αυτή την προσπάθεια συμφιλίωση του περιβάλλοντος με την οικονομία και βεβαίω το περιβάλλον μπορεί να στηρίξει την οικονομία. Ο κ. Φράνκο τα είπε αυτά. ορισμένε από τι διατυπώσει των τροπολογιών ίσω οδηγούν σε διαφορετική κατεύθυνση. Όταν μιλούμε για την εξασφάλιση ισορροπία μεταξύ οικονομική ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος τροπολογία 24 νομίζουμε ότι αυτό ίσως είναι ω διατύπωση λίγο επικίνδυνη διότι φαίνεται να προσπαθεί να αποκαταστήσει μια ισορροπία μεταξύ δύο διαφορετικών στοιχείων. Για την πολιτική των απορριμμάτων, αυτά τα είπε για λογαριασμό μου θα έλεγα ο κύριος Γκερμπραντή, πρέπει να προχωρήσουμε όντως οι τροπολογίες του εισηγητού μας επαναφέρουν λίγο στο status quo και για τις πρώτες σύλλες που διαθέτουμε. Δεν μπορούμε το 2020 να εξακολουθούμε να καίμε ε, πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν. Γι' αυτό και μας αρέσει η ιδέα της κυρίας Άουκεν και άλλων. Για τις τροπολογίες τώρα για την βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή συμφωνούμε με ορισμένες από αυτές τονίζουμε μία ανησυχία όταν μιλείτε για την ενίσχυση του πλαισίου, ε, νομικού πλαισίου. Εμείς θα θέλαμε να ενισχυθεί το σύνολο του νομικού πλαισίου και όχι μόνο αυτό για, για την βιώσιμη ανάπτυξη και παραγωγή μάλλον. Για την εφαρμογή, ε, ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τις ιδέες. Ορισμένα προβλήματα έχουμε για να δεχτούμε την ανάλυση της ε, τροπολογίας 46 που λέει ότι τα προγράμματα εφαρμογής εξαρτώνται από την περιπλοκότητα της ε, νομοθεσίας για το περιβάλλον και τις, και τις ε, συχνές αλλαγές της. Ελπίζουμε ότι δεν θα περιληφθεί τελικά στην τελική μορφή του προγράμματος. Για το Impel τώρα, εδώ μας ενισχύει λίγο με την έννοια ότι ορισμένες από τις τροπολογίες, παρόλο που δεχόμαστε την πρόθεσή τους, ίσως να μην είναι πολύ ρεαλιστικές. Το ΙΜΠΕΛ είναι ανεξάρτητο όργανο, δεν μπορούμε να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν. Κάνουν δύο peer reviews το χρόνο. Είναι μάλλον απίθανο να δεχθούν να κάνουν πολύ περισσότερα. Βέβαια πρέπει να εξασφαλίσουν και την χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα LIFE εκεί, επομένως πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας. Για τους στόχους ακόμη 6 και 9 για τις επιδοτήσεις. Πάλι συμφωνούμε με τα σχόλια του κυρίου Γκέρ Μπράντι, πρέπει να προχωρήσουμε. Μιλούμε για εντοπισμό των επιδοτήσεων μετά για την αφαίρεσή τους. Ο ΩΣΑ έχει προβλέψει καλούς ορισμούς και εμείς συμφωνούμε με αυτούς. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς προτεραιότητες τώρα, τμήματα του κειμένου έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Αυτό ισχύει η τροπολογία 70, Universal Membership of UNIP. Θα εκδώσει νέα ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διάφορες ιδέες για το εμπόριο και την αμοιβαιότητα. Σημειώνουμε την δέσμευση του εισηγητού να τηρήσουμε τους κανόνες του ΠΟΕ. Δεν είμαστε βεβαίες όμως ότι όλες αυτές οι τροπολογίες πραγματικά αποκρίνονται σε αυτή την δέσμευση. Ευχαριστώ. Κύριε Και υπάρχει και δεύτερος εισηγητής εμπειρογνώμων που έχει εργαστεί πολύ σκληρά στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τον ε, συναδελφό μας που είναι εμπειρογνώμων στα αγροτικά και τον παρακαλώ να λάβει το λόγο για δύο λεπτά. Γιατί κάνει σχετική έκθεση στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Γκρότε για την ευκαιρία που μου δίνετε. Όντως η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διεξάγεται σήμερα συζήτηση στην Ολομέλειά μας, δηλαδή έχουμε προχωρήσει με την έκθεσή μας. Δεν είναι βέβαια σύμπτωση το γεγονός ότι ε, βρισκόμαστε σε ένα έτος χωρίς πρόγραμμα δράσεως, διότι η Κομισιόν με τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και τις 7 ε, πρωτοβουλίες έχει δεσμευτεί από άψη περιβαλλοντική πολιτική. και εμείς αναρωτηθήκαμε αρχιτεκτονικά ας πούμε αυτό το 7ο πρόγραμμα δράσεων πώς εντάσσεται μέσα στο συνολικότερο πλαίσιο Χαιρόμαστε βέβαια καταρχήν για το πρόγραμμα δράσεων, το βρίσκουμε όμως πολύ περιορισμένα φιλόδοξο. Πολύ περιορισμένα φιλόδοξο και πολύ ε, ασαφές. Γι' αυτό προχωρούμε πιο έντονα, ας πούμε, πιο δραστικά και λέμε ότι μάλλον είναι έκθεση καταγραφής της κατάστασης του περιβάλλοντος και λιγότερο έγγραφο προθέσεων. Και ίσως μπορεί να ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα. Μέγα μέρο των προβλημάτων, όπω ελέγχθη, το γράφει και το πρόγραμμα, αλλά ελέγχθηκε ήδη, μέγα μέρο των προβλημάτων οφείλεται στο ότι οι χώρε μέλη αποτυγχάνουν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, διότι δεν έχουν επαρκή πολιτική βούληση. Τότε διαρωτώμεθα εμεί, αυτό το 7ο πρόγραμμα δράσεων δίνει απαντήσει για το πώ θα ασκηθεί κάποια πίεση στι χώρε μέλη. Και εμείς εδώ κάνουμε και μια διασύνδεση με την οικονομική κρίση. Επεξεργάζονται μηχανισμούς για την επιβολή κυρώσεων για την οικονομική κρίση. Κάτι παρόμοιο θα θέλαμε και στον τομέα του περιβάλλοντος. Ίσως μάλιστα να μπορεί να τεθεί το ερώτημα, από την πλευρά σας δηλαδή, εάν μεταξύ αυτών των νέων προτεραιοτήτων, αν δηλαδή αυτές οι νέες προτεραιότητες είναι πραγματικά σωστά επιλεγμένες. Τα είπε ο κ. Φλόρεντς, είναι οι μεγάλες προτεραιότητες της πολιτικής του κλίματος, αλλά αυτό δεν αναφέρεται τόσο πολύ. Πιο πολύ αναφέρεται το αστικό περιβάλλον. Τι είδους στάθμιση είναι αυτή. Εμείς λοιπόν έχουμε ιδιαίτερα κριτική στάση και ασφαλώς είμαστε στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε με τον εισηγητή σας ή και τους κοιόδη εισηγητή σας. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σα και τον σκιωδη εισηγητη σα. είναι επίσης παρούσα σήμερα, όπως άλλωστε το πράττει συχνά στην Επιτροπή μα, και γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ε, μία από τις κύριες προτεραιότητες της για το εξάμεινό της. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω. Η το σχέδιο αυτό, το πρόγραμμα αυτό είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα της Ελλανδικής Προεδρίας σε θέματα περιβάλλοντος. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τον κύριο Φράγκο και την ομάδα του. Και βέβαια και με τον κύριο Λάινεν είχαμε πολύ σημαντική συνεργασία στην προηγούμενη έκθεση. Στο Συμβούλιο έχουμε οκτώ ομάδες εργασία που έχουν συγκληθεί τους τελευταίους τρεις μήνες και άλλες πέντε ομάδες θα ολοκληρωθούν πριν το στις αρχές Μαρτίου. 52 διμερείς επίσης έχουν λάβει χώρα με τα κράτη-μέλη. Ως αποτέλεσμα το κείμενο έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο Συμβούλιο. Θέλουμε να πετύχουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ακούσαμε την συζήτηση στην Επιτροπή σας τον περασμένο μήνα και μαζί με την σημερινή συνεδρίαση χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την έμφαση που δείτε στην εφαρμογή και για την ποιότητα των συζητήσεων. Η Ιρλανδία έχει αντιμετωπίσει σημαντικέ δυσκολίε στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουμε θετικέ ε, εμπειρίε ακολουθώντα την προσέγγιση τη Κομισιόν. Ω αποτέλεσμα, οι ανοιχτέ ε, διαδικασίε επί παραβάση έχουν μειωθεί από 32 2010 σε 12 σήμερα ε, και νομίζουμε θα κλείσουν και άλλε τρει τον επόμενο μήνα προσεγγίσεις όπως οι συμφωνίες εφαρμογή, εταιρικές συμφωνίες εφαρμογής και άλλες ήταν πολύ επιτυχή στην Ιρλανδία και σας τη συστήνω. Ε, καλωσορίζουμε την έκθεσή του εισηγητή και ιδιαίτερα την ενίσχυση της γλώσσα σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Αυτό το έχει λάβει υπόψη του και το Συμβούλιο. Ε, διαβάζουμε το κείμενο σε ό,τι αφορά την, το στόχο προτεραιότητα 9 ε, και αναθεωρούμε το κείμενο έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη ε, οι τελευταίε εξελίξεις στο πρώο περιβάλλον του ΟΗΕ το, του Ναϊρόμπι στι αρχές του έτου. Ε, θέλουμε να συμφιλώσουμε τι ε, φιλοδοξίε ε, διαφόρων κρατών μελών σε ό,τι αφορά το έδαφος για να αποφύγουμε ε, μια μειοψηφία που θα μπλοκάρει το κείμενο. Ας αρχίσουμε με το τι θέλουμε να κάνουμε για τα εδάφη μας στην Ευρώπη. Συνολικά λοιπόν, Πρόεδρε, πιστεύω ότι ευθυγραμμίζεται αρκετά το κείμενο του Συμβουλίου με την ε, θέση της έκθεση του εισηγητή. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία, να πω ότι ευχαριστούμε την Κομισιόν που υπέβαλε το κείμενο τόσο σύντομα. Ε, είναι πολύ σημαντικό να υιοθετηθεί το συντομότερο διότι υπάρχει κενό ανάμεσα στο έκτο και το έβδομο πρόγραμμα. Μα χαροποιεί ιδιαίτερα το format ε, και ο τρόπος παρουσίασης ε, της έκθεσης κομισιών. Ε, Επίση, το χρονοδιάγραμμα τη Επιτροπή σα μα ικανοποιεί. Ε, δεδομένου μάλιστα ότι τα δύο όργανα κινούνται προ την ίδια κατεύθυνση ό,τι αφορά το περιεχόμενο, περιμένουμε ότι η πρώτη ανάγνωση θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Limes, for your statement. So, now last but not least, the rapporteur, Mr. Franco. Ο κύριος Φρανκο, ο εισηγητής. Δεν είχαμε πρόθεση να αποδυναμώσουμε το κείμενο. Ε, άκουσα με μεγάλη προσοχή και τους συναδέλφους και κάναμε και μία ε, παρουσίαση μαζί με την ΕΟΚΕ για, την, για το πρασίνισμα της ΚΑΠ. Στην Ολομέλεια χρειάστηκε να διευθετηθεί και να ψηφιστεί αυτό το θέμα για, για τα δάση και τα δασοκομεία. Είχα ε, αναφερθεί, θα ήθελα να πω και παράλληλα και στις θάλασσες και τους ωκεανούς και τα κείμενα από τη Δευτέρα είναι διαθέσιμα και ε, στα αγγλικά, αν ε, και σήμερα είναι η μέρα των γαλλόφωνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, τα οποία θα λάβω υπόψη πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ κύριε Φράγκο. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών 25 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 24 Απριλίου και στην Ολομέλεια πιθανότατα θα καταλήξει ε, στον ε, μήνα Ιούνιο, έκτο δηλαδή. Ευχαριστώ για την συζήτηση και προχωρώ στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι ο στόχος μείωσης των εκπομπών από τα επιβατικά αυτοκίνητα με εισηγητή τον κύριο Ούλμερ που λαμβάνει για 5 λεπτά τον λόγο. Μας μένει ακριβώς μια ώρα. Ήδη, ήδη πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτα θα ήθελα να παρακαλέσω οι σχετικές συνομιλίες να γίνουν έξω από την αίθουσα, όποιοι επιθυμούν δηλαδή, ώστε να μπορέσει ο κύριος Ούλμερ να κάνει την παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις και τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει και είναι περίπου 200 τον αριθμό. Αποκρισταλώνονται βεβαίως μέσα από αυτές διάφορα θέματα όπου φαίνεται να μπορούν να ε, προκύψουν και συμβιβασμοί για την επίτευξη πολλών από τους στόχους. Πρώτα, ο μακροπρόθεσμος στόχος που διαφαίνεται είναι μεταξύ 2014 και 2017 ένα στόχος 50 έως 80 γραμμαρίων νομίζω ότι θα πρέπει να περιλάβουμε και ισοδύναμα του διοξιδίου του άνθρακος και να δούμε προς ποια τεχνολογική κατεύθυνση θα προχωρήσει το μέλλον του αυτοκινήτου. για να περιληφθούν και άλλοι τρόποι κίνησης, για παράδειγμα ηλεκτρική ενέργεια κλπ. Δεύτερο, εν προκειμένου, είναι τα λεγόμενα super credit, φαίνεται να μπορούμε να δώσουμε super credit της τάξης των 2-4 γραμμαρίων ανά Και αυτές να μπορούν να πιστώνονται. Εάν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν βέβαια από το 2020 και μετά μπορεί να λήξει η προσπάθεια αυτή. Ο περιορισμός του συμψηφισμού βέβαια θα πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον, δεν, εφόσον ε, ε, ορισμένα όρια. Δηλαδή αν φτάσουν στα 50 γραμμάρια ή αν ληφθεί ως μέτρο το 50%. Επομένως οι εκπομπές να είναι στα 60 70 γραμμάρια. ορισμένα αυτοκίνητα θα εκπίπτουν του συστήματο αυτού. Αυτό σημαίνει ότι αν μπορούν να είναι οι πιστώσει των μορίων αυτών μεταξύ 16 και 20 ώστε να μειωθεί η καμπύλη μεταξύ 2016-2023 ώστε να αποτελέσει ευνοϊκό κίνητρο για να βγουν νέα επιβατικά αυτοκίνητα στο, στην αγορά. Το τρίτο που πρέπει να συζητήσουμε είναι ο κύκλος δοκιμασιών. Ασφαλώς και θα πρέπει να εισαχθεί νέος κύκλος δοκιμασιών και για την προστασία των καταναλωτών αλλά και να επιτρέπει και συγκρισιμότητα με τις πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες. Το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος παγκόσμιας ισχύος κύκλος δοκιμασιών που να επιτρέπει την σύγκριση των διαφόρων μοντέλων με περιορισμό της ε, γραφειοκρατίας Που βέβαια εξυπηρετεί και τους καταναλωτές σε όλες τις χώρες. Αυτό για την ώρα φαίνεται να είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή υπάρξει ο κύκλος δοκιμασιών, μπορεί αυτό να γίνει ανα πάσα στιγμή το παγκόσμιο δηλαδή σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει και μια συγκρισιμότητα με τον ενισχύοντα στόχο των 95 γραμμαρίων. Πολλέ τροπολογίες έχουν κατατεθεί για τις οικολογικές καινοτομίε, Εκεί εγώ φαντάζομαι να μπορεί να υπάρξει μια πολύ απλή έγκριση με στόχο ίσως το ένα γραμμάριο. Μέχρι τώρα υπάρχει μόνο μια οικολογική καινοτομία από ένα γερμανό κατασκευαστή. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες έχουν απορριφθεί. Είναι πολύ γραφειοκρατικές και δαπανηρές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μέσα σε δύο η τρεις μήνες η Κομισιόν να μπορεί να χορηγεί έγκριση και όχι μέσα σε ε, ακαθόριστο χρονικό διάστημα. διάστημα. Το άλλο θέμα είναι το θέμα του ίχνους που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ για την εκπομπή διοξιδίων του άνθρακος. Αυτό το footprint εμένα δεν μου φαίνεται ενδεδειγμένο. Γιατί ρόλο παίζουν εδώ οι διαστάσεις του αυτοκινήτου αλλά και το βάρος. διότι τότε θα σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορεί να εκλείει περισσότερο διοξίδιο του άνθρακος. Το μακρύτερο ή φαρδύτερο αυτοκίνητο σημαίνει βεβαίως ότι καταναλώνει το αυτοκίνητο και μεγαλύτερη ε, επιφάνεια. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερα πάρκινγκ ε, ε, παίρνει περισσότερο χώρο πάνω στο δρόμο, άρα περισσότερες κυκλοφοριακές εχμές και ούτω καθεξής. Μείωση της μάζας, ωστόσο, θα οδηγήσει το αυτοκινήτο δηλαδή και σε μείωση της ε, εκπομπής οξυδίου του άνθρακος. Αυτό ο δρόμο μου φαίνεται ορθότερος. Και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι σε όλο τον κόσμο εκτό από τις ΗΠΑ. Εν τέλει θέλω να δηλώσω ότι τον Απρίλιο προβλέπουμε δύο συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών όπου θα προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε κοινέ συμβαστικέ προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ούλμερ. Ακολουθούν οι σκιώδεις εισηγητές και θα σας διαβάσω τα ονόματα. Έχουν επίσης δει στο λόγο und Anna Rosbach. Habe ich noch jemanden vergessen? ξέχασα κανένα όνομα. Μάλιστα, η κυρία Ρόσπαχα αντικαστά τον κύριο Κέραναν. Θα παρακαλέσω τις και τους συναδέλφους να περιοριστούν στα γνωστά δύο λεπτά. Μάριο Πυρίλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι τροπολογίες των συναδέλφων επιβεβαιώνουν το στόχο των 95 ε, γραμμαρίων ε, διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο μέχρι το 2020. Έτσι, αυτή το βιομηχανία της Ευρώπης θα πρέπει να προγραμματίσει τη δραστηριότητά της μέχρι τότε. Όσον αφορά τα, το σύστημα των ε, υπερμορίων, οι θέσεις διαφέρουν. Εγώ προσπάθησα να φτάσω σε ένα γεφύρωμα των 95 γραμμαρίων ε, με άλλες προτάσεις. Εγώ είμαι υπέρ μιας θετικής ε, βαθμολόγησης τη στιγμή που μπορούν να πολιθούν ε, και οχήματα τα οποία ε, αφορούν και εκπομπές μέχρι 35 γραμμάρια. Μιλάμε για πώληση 20.000 οχημάτων και δέχομαι και τις τροπολογίες των άλλων συναδέλφων. Δεν ξέρω κατά πόσο ο στόχος των 95 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο μέχρι το 2020 θα μπορούσε να ενταχθεί μέχρι τον κύκλο 2020. Θα πρέπει να ξαναδούμε τον κύκλο ε, δοκιμών έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο αντικατοπτρίζει τους νέους κανόνες περιοδήγησης οχημάτων και πολλές φορές οι καταναλωτές ε, δεν έχουν πραγματικές πληροφορίες για τις πραγματικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό θεωρώ μέχρι το 2014 ότι θα πρέπει να ορίσουμε τον παγκόσμιο κύκλο δοκιμών που θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2017. Εάν αυτό τεχνικός δεν είναι δυνατόν, η Επιτροπή θα πρέπει να δεχτεί μία μεταβατική φάση αλλάζοντας τον ενισχύει κανονισμό. Τέλος, ως προς τους στόχους μετά το 2020, η παρούσα τεχνολογία δεν να προβλέψει πραγματική μείωση του στόχου των 95 γραμμαρίων. Γι' αυτό δεν έχει νόημα να ορίσουμε νέο στόχο. Αντίθετα θα πρέπει να δώσουμε ποσοτικά στοιχεία μεταξύ 60 και 65 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο ε, ανάλογα με τις μελέτες αντικτύπου που θα έχουν γίνει μέχρι τότε με βάση τα νέα οχήματα τα οποία θα κατασκευαστούν. Chris Davis. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες βελτίωσης ε, των συνάδελφων της Επιτροπής Βιομηχανίας. Όταν συζητήσαμε την νομοθεσία το 2008, είδαμε μια βελτίωση 50% στον αριθμό των χιλιόμετρων ανά λίτρο βενζίνης ή δίζελ ε, των ε, νέων αυτοκινήτων από το 2008 και μετά. Αυτό είναι πολύ καλό νέο για τους πολίτες μας και για το περιβάλλον. Γιατί αυτό βέβαια σημαίνει και μείωση κατά 50% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Σημαντική μείωση. Στην ε, συνάντηση με τους ε, κατασκευαστές ανταλλακτικών μας είπαν ότι τα δύο τρίτα αυτής της βελτίωσης ε, προέκυψαν ως αποτέλεσμα νομοθεσίας. Συνεπώς η καινοτομία υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή από τις απαιτήσει που ε, επιβάλλουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία περνάει πολύ δύσκολε στιγμές με χαμηλή ζήτηση και υπερβάλλουσα παραγωγή. Κάπως θα πρέπει να λυθεί το θέμα, αλλά αν δεν συνεχίσουμε να καινοτομούμε όπως κάναμε τα τελευταία χρόνια ε, δεν θα επιβιώσουμε, θα, η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη. Ε, όταν επανέλθει η οικονομική ανάκαμψη κάποια στιγμή. Επιβεβαιώνω το στόχο των 95 γραμμαρίων. Ε, υποστηρίζω ένα βαθμό super credits για να προωθήσουμε την καινοτομία πολύ χαμηλής κατανάλωσης διοξιδίου του άνθρακα θέλουμε ένα στόχο, μακροπρόθεσμο στόχο του 2025, ε, υπό αναθεώρηση βέβαια, ενδεικτικό στόχο. Θέλουμε επίσης οι δοκιμές, ο κύκλος δοκιμών να γίνει πιο αυστηρός, έτσι ώστε να αποφεύγουμε ε, τις παραβιάσεις που μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή. Ε, μιλήσαμε για τις οικολογικές κοινοτομίες. Εγώ ήμουν πολύ επικριτικός όταν υιοθετήθηκε καταρχήν νομοθεσία. Εγώ θεωρούσα ότι η οικολογική καινοτομία ε, θα θεωρείται ως πιο αδύναμος κρίκος. Στην πραγματικότητα ήταν, έγινε με πολύ αυστηρή εφαρμογή νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά το οικολογικό ίχνος, ε, σε προηγούμενο νομοθετικό κείμενο είχαμε πει ότι θα μπορούσε να ακολουθεί, θα μπορούσε να ακολουθεί είτε το, η προσέγγιση του ίχνους είτε η προσέγγιση της μάζας. Ε, οι Αμερικανοί αν θέλουν, αν θέλουν σοβαρά να διαπραγματευτούν μια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα εμπλέξουν σίγουρα το ίχνος, το οικολογικό ίχνος, ε, οπότε ας το έχουμε υπόψη μας. Ε, χαίρομαι που ε, ο κ. Σολμέρ ε, είναι δεκτικό σε προτάσεις. Θα δουλέψουμε μαζί του με πολύ ενθουσιασμό. Very much. Chris, Ja, vielen äh, Χάρμς, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έρχεται και πανέρχεται, Η ρύθμιση δηλαδή τη εκπομπή διοξιδίων του άνθρακο από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Για λογαριασμό τη ομάδα μου, έχω, βάλει, έχω υποθε... καταθέσει μια τροπολογία για την μέση τιμή εκπομπή του 2020, όπου θεωρούμε ότι το impact assessment της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι, 25, ε, ότι, ότι είναι δυνατόν, είναι εφικτό όριο 25 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο και ότι το σχετικό υψηλότερο κόστος των αυτοκινήτων θα αντισταθμιστεί από την εξοικονόμηση καυσίμου. Βέβαια γνωρίζω ότι βρίσκομαι σε θέση μειονότητα εν προκειμένου. Αλλά, επαναλαμβάνω, η μελέτη αντικτύπου Impact Assessment τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα λέει αυτά τα πράγματα και πρέπει να ληφθεί. 95 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, προφανώς, από την άποψη της προστασίας των καταναλωτών, δηλαδή οικονομικά αυτοκίνητα, ε, δεν είναι βέβαια και το καλύτερο, μπορεί να βελτιωθεί ήδη από το 2020. Για το 2025 καταθέτουμε τροπολογία με πιο φιλόδοξο στόχο, τα 60 γραμμάρια δηλαδή διοξιδίου του άνθρακος ανά χιλιόμετρο. Νομίζουμε ότι βάζοντας πλέον φιλόδοξους στόχους μπορεί να επιτύχει κανείς περισσότερη και καλύτερη καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω πρόθεσμα. Καλύτερα έτσι παρά να προχωρεί αργά και διστακτικά. Για τα λεγόμενα super credit, κατά τη γνώμη μου δεν χρειαζόμαστε τέτοια υπερμόρια. Και μετά το 2020 η αγορά του αυτοκινήτου θα κυριαρχείται από τις συμβατικές μορφές προώθησης ενέργειας δηλαδή. Γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται φιλόδοξη επιβολή των στόχων που συμφωνούμε και να μην αφήσουμε παραθυράκια ανοιχτά στην ομοθεσία με τα λεγόμενα super credit που αναλόγως του πώς εφαρμόζονται μπορούν να οδηγήσουν σημαντικά στην αποδυνάμωση των στόχων. Και θεωρώ ότι μεταξύ ημών των σκιωδών εισηγητών πρέπει να επανεξετάσουμε τις τροπολογίες, διότι ορισμένες από αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατά 20% μικρότερη εξοικονόμηση στις συμβατικές ενέργειες. Τέλος, κύκλος δοκιμασιών, υπάρχει καλός τέτοιος κύκλος δοκιμασιών. Ε, κύριε Πρόεδρε, και οι άλλοι μίλησαν παραπάνω από δύο λεπτά. Συγγνώμη, ο κύκλος δοκιμασιών μπορεί λοιπόν να εισαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίω σε ό,τι αφορά την προστασία καταναλωτών είναι στα λόγια και αυτά που κάνουμε με τον κύκλο δοκιμασιών είναι πραγματική εξαπάτηση των καταναλωτών η κυρία Άννα Ρόσπαχ που αντικαθιστά τον κύριο Κάλαναν. Ευχαριστώ, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια στα αγγλικά. Ως προς το στόχο θεωρούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, από 130 ε, περνάει για το 2015 και 95 γραμμάρια μέχρι το 2020. Είναι πολύ φιλόδοξη η στόχη, αλλά η βιομηχανία θεωρεί ότι είναι σχετικά ε, βιώσιμη. Δεχόμαστε το, τη θέση του εισηγητή να δεχτούμε τη διπλή εξαίρεση και να δοθούν πριν στους ε, μικρούς κατασκευαστές. Απορρίπτουμε τις ε, τροπολογίες που ε, δεν δέχονται την ε, μείωση του άχθους για τις μικρές βιομηχανίες μέχρι το 2020. Πολλοί μίλησαν για αλλαγή χρήσης, μιλάμε δηλαδή για αλλαγή από το αποτύπωμα στη μάζα και αυτό θα πρέπει να το δούμε στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα μας διέπει το 2020 σε σχέση με τη διαδικασία δοκιμών. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτός, αυτή η παγκόσμια διαδικασία δοκιμών ελαφρών δοκιμάτων, οχημάτων συγχωρείτε, και θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη τα οικονομικά δεδομένα. Δεν θα πρέπει εσπευσμένα να ε, θέσουμε μία νέα διαδικασία η οποία θα μπορούσε να υποβαθμίσει το στόχο του 2020. Ευχαριστούμε την ανά Φλόρεντς. Ευχαριστώ τον Τόμας Ούλμερ και χαίρομαι που δηλώνει διατεθειμένος να συμφωνεί σε συμβασμούς. Δεν θα μπω καν σε όλα αυτά τα θέματα του ενός γραμμαρίου παραπάνω ή παρακάτω. Αν σκεφτεί κανείς τι αυστηρούς κανόνες έχει επιβάλει στην αυτοκινητοβιομηχανία η Κομισιόν με τα ETS κλπ. Και μετά έρθει και δει πόσο αδύναμη είναι τούτη εδώ η οδηγία. Διαρωτώ με τι κριτήρια εφαρμόζει η Κομισιόν και ιδίω η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Η αυτοκινητοβιομηχανία καλείται να μειώνει τα διοξίδια του άνθρακα κατά 1,7% τον χρόνο είναι μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα. Η Κομισιόν θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι πλέον φιλόδοξη. Λυπούμε πολύ. Ένα άλλο μέγα θέμα είναι ο κύκλος δοκιμασιών. Αγαπητή Κομισιόν, ποιον περιμένετε. Θέλετε να εγκαταλείψετε το θέμα στην Ευρώπη και να περιμένετε τον παγκόσμιο κύκλο δοκιμασιών. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταθέσουμε καλές προτάσεις αύριο, μεθαύριο, εσείς είστε ο, ο των συνθήκων, να πιέσετε λίγο και την αυτοκινητοβιομηχανία. Μπορούμε να επωφεληθούμε πολύ περισσότερη ειλικρίνεια. Έχετε, έχουν δει και ορισμένες ε, συνάδελφοι που είπαν ότι εξαπατούμε τον κόσμο με αυτούς τους κύκλους δοκιμασιών. Ασφαλώς και πρέπει να επιβάλλουμε άλλους κανόνες. Να είμαστε και ρεαλιστές, αλλά πράγματα αυτά να είναι εφικτά είμαι και διατεθειμένος να συμφωνήσω με τον Τόμας Ούλμερ για τα κριτήρια που θα πρέπει να είναι ωστόσο συγκρίσιμα. Αλλά αγαπητοί Κομισιόν, να καταβάνετε κάποια μεγαλύτερη προσπάθεια, όχι απαραίτητα στα γραμμάρια, αλλά στην καινοτομία. Αυτά τα γράφετε και τα ξαναγράφετε. Χρειαζόμαστε καινοτομία. Ναι, αλλά εσείς δεν έχετε υποβάλει κριτήρια για την καινοτομία. Ευχαριστώ. Καρλ Χάιντς, Κορίν Λεπάζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που με αυτή τη συζήτηση μας δίνει τη δυνατότητα να βρούμε σωστές ε, τροπολογίες. Θα ήθελα να επανέλθω ως προς την ανάγκη να έχουμε έναν ευρύ ορίζοντα για την ε, ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Θα πρέπει να συμφιλιώσουμε ε, το περιβάλλον με τα συμφέροντα του καταναλωτή και της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στόχους και μετά το 2020 και φιλόδοξους στόχους γενικότερα. Εγώ μιλώ για 60 γραμμάρια διοξίδιου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο σε μια τροπολογία. Νομίζω ότι τα υπερμόρια ενέχουν και κινδύνους, διότι αποδυναμώνουν τους στόχους ε, τα όρια εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα ως προς τις δοκιμές. Θα πρέπει να τις ξαναδούμε και αυτό το ταχύτερο δυνατόν διότι το ε, παρόν σύστημα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και Πολλές φορές τα οχήματα δεν αντικατοπτρίζουν τις προδιαγραφές που αρχικά προτείνονται. Θα πρέπει να ορίσουμε έναν φιλόδοξο στόχο και έτσι θα ε, μειώνονταν οι εκπομπές και τα καύσιμα και αν χρησιμοποιήσουμε τη μάζα ως κριτήριο δεν θα έχουμε ελαφρύτερα οχήματα. Γι' αυτό ίσως θα ήταν ε, σκόπιμο να μιλάμε για το αποτύπωμα και όχι το κριτήριο της μάζας. Ευχαριστώ. Λάινεν. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Νομίζω ότι τα πράγματα ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά. Φαίνεται που μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια πλατιά πλειοψηφία καταρχήν στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια. Τα 95 γραμμάρια για το 2020 νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένας ε, ε, στόχος ε, ένα πρώτος στόχος, θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε βέβαια, αλλά δεν πρέπει να αλλάζουμε τους κανόνες στο μέσο του παιχνιδιού. Αφού πετύχουμε τα 95 γραμμάρια, σίγουρα θα έχει δημιουργηθεί και μια ορμή ο Μάριο Περίλο έκανε ε, πρόταση να ε, μην έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο αλλά ε, μια ψαλίδα, μια και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή τι θα, πώς θα πάει η τεχνολογία. super credits, εγώ θα έλεγα ότι δεν τα χρειαζόμαστε, αλλά τα εισάγουμε θα πρέπει να περιοριστούν σε ε, δύο γραμμάρια για παράδειγμα όπως πρότειναν πολλοί. Από ό,τι χρειάζεται η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται κίνητρα για να διαθέσει καινούργια αυτοκίνητα στην αγορά. Αν αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με τις υπερπιστώσεις ε, τότε ε, θα το δούμε. Είμαι λοιπόν υπέρ ενό ε, περιορισμού σε αυτό το εργαλείο. Ε, το, ο κύκλος των δοκιμών θα πρέπει επίσης να γίνει πιο αυστηρός σε ό,τι δεν αφορά ε, το ίχνος έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες για ηλεκτρικά ή αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα υδρογόνου δεν μπορούμε να εργαστούμε από τη βάση εκπομπών διότι δεν υπάρχουν εκπομπές συνεπώς θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει με αυτά τα οχήματα, ηλεκτροκίνητα, οχήματα ή οχήματα που κινούνται με υδρογόνο. Τα Η Κομισιόν θα πρέπει να δει το θέμα αυτό του ίχνους, ε, της αξιολόγησης ε, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Είναι προφανές ότι αν χρησιμοποιήσουμε τις... το, το ίχνος θα έχουμε ε, λιγότερες ε, ε, επιπτώσεις από τη μάζα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λάινεν. Ε, πέντε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα έχει φτάσει η κατανάλωση ως με ένα αυτοκίνητο μεταξύ αυτών και το δικό μου. Ε, αν κινείστε με 120-130 χιλιόμετρα την ώρα στο Βέλγιο, την Ολλανδία, με ένα σχετικό καινούριο, σχετικά καινούριο αυτοκίνητο, ε, ε, όμως ε, δεν, ε, η κατανάλωση δεν πέφτει κάτω από τα 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα συνήθως. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. διότι άλλο το τι λέει το manual, μπορεί να λέει 5, και άλλο τι γίνεται στην πραγματική ζωή, που τελικά το 5 γίνεται 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ο κύκλος δοκιμών θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματική ε, χρήση. Ε, το αν αυτό θα γίνει παγκοσμίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το δούμε, αλλά αν θέλουμε να ε, κινητοποιήσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία προστατεύοντας το περιβάλλον, χρειαζόμαστε και φορολογικά κίνητρα. Και όταν έχουμε πολύ περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πρέπει να δούμε πώς θα ενταχθούν σε όλο αυτό το σύστημα. Η φορολόγηση των αυτοκινήτων θα πρέπει να εναρμονιστεί στην Ευρώπη κατά την άποψή μου. Χρειαζόμαστε τα καλύτερα δυνατά προγράμματα, χρειαζόμαστε ε, ένα... Ε, ε, χρειαζόμαστε και το φορολογικό σύστημα να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός, διότι ε, οι άνθρωποι πραγματικά αντιδρούν σε κίνητα και αντικίνητρα φορολογικής φύσης. Και στην τρέχουσα νομοθεσία έχουμε τα super credit. Εγώ τα υποστήριξα τα super credit διότι θεώρησα ότι με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε το δυνατόν συντομότερο εναλλακτικέ πηγές ενέργειας για τα αυτοκίνητα εφόσον δηλαδή η περιγραφή είναι ουδέτερη. Ωστόσο είμαστε ακόμα μακριά από το στόχο αυτό. Ζήτησα λοιπόν ρύθμιση των ε, υπερμορίων αυτών με τρόπο που ε, ναι μεν να προσφέρουν επιβράβευση όσων εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή, να μην υπονομεύσουν όμως από την άλλη μεριά το όριο των 95 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο που νομίζω σας βρίσκει όλους και όλες σύμφωνους στη συζήτηση αυτή. Αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον, ο κύριος Ούλμερ άνοιξε την αγκαλιά του σήμερα, μας προσφέρει τη δυνατότητα ε, συμβασμών και η Επιτροπή Βιομηχανίας ψήφισε χθε νομίζω ότι κινείται προς την κατεύθυνση την δική μας. Έχω ωστόσο ακόμη μία συνάδελφο που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, αν επιθυμεί κάποιος ακόμη. Αλλιώς έχετε το λόγο. Βέβαια, κοιτάξτε λίγο και το ρολόι. Κύριε Μέρκες, ε, χτες ψηφίσαμε στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Περίμενα η Επιτροπή Περιβάλλοντος να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένη σε ένα αρισμό θεμάτων, για παράδειγμα δοκιμές, η Επιτροπή Κομισιόν ε, αποδέχεται ότι η διαχείριση των κύκλου δοκιμών ε, δεν είναι σωστή Αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες επιλογής ε, όταν η αυτοκινητοβιομηχανία κάνει τους, ε, τις δοκιμές. Από την άλλη μεριά τίθεται και το θέμα του ποιος θα κάνει την, παρακολου... <coughs> Συγγνώμη, την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το θέμα των super credits, Μερικέ φορέ χρειάζονται περισσότερη προσαρμογή στην πραγματικότητα διότι δεν λειτουργούν πάντοτε. Εγώ πρότεινα να έχουμε ένα ε, κριτήριο σύγκρισης που θα λαμβάνει υπόψη το μέσο όρο στην αγορά. Οπότε ανάλογα με το αν η τιμή είναι πάνω ή κάτω από αυτό το όριο, το benchmark, ε, θα υπάρχει ένα σύστημα ε, κύρωσης, κυρώσεων ή ανταμοιβών. Αυτή τη στιγμή ε, τα super credits δεν είναι αρκετά ευέλικτα. Δεν είναι ευέλικτο σύστημα. Γιατί, γιατί η αγορά μεταβάλλεται. Μην βλέπετε ότι γίνονται διαδηλώσει σε ό,τι αφορά την, το μέλλον τη αυτοκινητοβιομηχανία. Α είμαστε προσεκτικοί. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Θα είμαι σύντομος. Διεξήχθη συζήτηση για μακροπρόθεσμους στόχους. Εδώ είναι σωστό να σημειωθεί η ωφέλεια που έχει προκύψει από τον στόχο των 95 γραμμαρίων. Έχει βοηθήσει την αυτοκινητοβιομηχανία και να σχεδιάσει και να καινοτομήσει. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και δείχνει την σημασία μακροπρόθεσμων στόχων, αλλά την σημασία επίσης της ασφάλειας σχεδιασμού για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να πιστοθεί με τη μείωση 3% που βλέπουμε στους κύκλους δοκιμασιών. Για τα super credit η Κομισιόν έχει διανύμει ένα μη έγγραφο για να, όπου συζητεί τις διάφορες παραλλαγές των super credit. Νομίζουμε ότι το banking είναι άσχημη ιδέα και το καθεστώς super credit μπορεί να προσφέρει κάποια κίνητρα βέβαια για την διάθεση στην αγορά αυτοκινήτων με πολύ χαμηλές εκπομπές καυσαρίων, αλλά πρέπει να έχει συγκεκριμένα κατόφλια και συγκεκριμένους περιορισμούς σε ό,τι αφορά το ποσοστό που μπορεί να υπονομεύσει εν τέλει τον στόχο. Το non-paper λοιπόν είναι σαφές για τις απαιτήσει αυτές όσον αφορά τον κύκλο δοκιμασιών και εκεί έχουμε κυκλοφορήσει σχετικό μη έγγραφο που δείχνει ότι η Κομισιόν προχωρεί σε βελτιώσεις για τον κύκλο δοκιμασιών. Προβλέπουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί κάτι σχετικό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το 2014. Δεν βλέπουμε λόγο να καθυστερήσει η βελτίωση αυτή, η οποία όντω θα βελτιώσει τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι καταναλωτές θα βελτιώσει την ακρίβεια των διαδικασιών δοκιμασιών και πολλοί από εσά τονίσατε ότι αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες αυτές δεν είναι άριστες. Μιλήσατε και για την οικολογική καινοτομία. Έχουν γίνει τέσσερι, έχουν προωθεί τέσσερις αιτήσει για Eco Innovation. Η μία ε, εγκρίθηκε, οι άλλες τρεις εξετάζονται. Νομίζουμε ότι λειτουργούν, αποδίδουν οι διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά διεξήχθη διαβούλευση με τους αρμόδιους stakeholders σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι διαδικασίες αυτές. Και καλύτερα να μην το οθήξουμε περισσότερο για τη λειτουργία διαδικασία. Κάποια άλλα σχόλια που ακούστηκαν για αξιολόγηση του κύκλου ε, ζωής, επίσης ε, του ίχνους και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων Έχουμε διάφορες μελέτες που βρίσκονται, στην, ε, βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές μακροπρόθεσμα. Ορισμένες θα δημοσιευτούν σύντομα, άλλες ε, θα έρθουν αργότερα, αλλά βρίσκουμε ότι είναι σωστό για τους μακροπρόθεσμους στόχους να περιμένουμε τα πορίσματα των μελετών αυτών. Ευχαριστώ και τέλος, λέει ο Πρόεδρος, ο Κύριε Ούλμερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τους κύκλους δοκιμασιών. Καλά θα ήταν η Κομισιόν να καταβάλει προσπάθεια ώστε οι προτάσεις που θα κάνει να μπορούν να έχουν και παγκόσμια ισχύ. Δεν βοηθεί πολύ μια αυτοκινητοβιομηχανία να χρειάζεται να προβλέπει ε, για κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστό βιβλιάριο με τις τιμές ανά κύκλο δοκιμασιών και ανά χώρα ή ήπειρο και ούτω καθεξής. Γιατί φαίνεται σαν η αυτοκινητοβιομηχανία να προσπαθεί να εξαπατήσει τους καταναλωτές. Δεν συμβαίνει αυτό. Χρησιμοποιεί η αυτοκινητοβιομηχανία τις δυνατότητες που τους προσφέρει ο νομοθέτης. η μείωση από 130 γραμμάρια σε 95 γραμμάρια μέσα σε μια πενταετία είναι ασφαλώς πολύ περισσότερο από 1,7% των χρόνων. Μπορούμε για τα υπερμόρια να ακολουθήσουμε μια κοινή γραμμή για να πούμε το 2020 έως 2025 θέλουμε φιλόδοξο στόχο αλλά προτιμούμε ένα είδος διαδρόμου παρά συγκεκριμένους αριθμούς και να καθορίσουμε από κοινού, αν δηλαδή θα μετράτε μόνο το διοξείδιο του άνθρακος ή πρέπει να μετρώνται και άλλες παράμετροι. Θα πρέπει να αναμένουμε ωστόσο τις αξιολογήσεις γιατί life cycle assessment σημαίνει 20 έως 30% του συνολικού διοξειδίου του άνθρακος που χρησιμοποιείται, μάλλον που ε, εκπέμπεται για την κατασκευή του αυτοκινήτου είναι και αυτό ένα από τα κέρια κριτήρια. Τι είστε και το ερώτημα αυτό μήπως πρέπει να επεκταθεί σε, στο να περιλάβει όλα τα αέρια που είναι επιβαρυντικά του κλίματος. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει ο στόχος, δεν θα αλλάξουν τα υπερμόρια, θα γίνουν δηλαδή όσο γίνεται πιο απλά, και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τι επόμενε συζητήσει με τους κύριου συζητητέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά, λέει ο Πρόεδρος. Λίγη εδώ η συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα την ξαναδούμε στις 24-25 Απριλίου, όπου θα γίνει η ψηφοφορία για, τις σημαντικές αυτές, για τη σημαντική αυτή έκθεση, διότι εδώ ασκούμε και βιομηχανική πολιτική αλλά και περιβαλλοντική πολιτική. Κάπου λοιπόν αυτά πρέπει να εξισορροπούνται με ευφύ τρόπο. Διότι πρόκειται βέβαια και για πάρα πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και η προστασία του καταναλωτού παίζει ένα σημαντικό ρόλο, καθώς και η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος και εν τέλει η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα και κλίματος αλλά και βιομηχανικής πολιτικής. Βέβαια δεν είναι μονάχα ε, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ε, ενδιαφέρει και το μείγμα ενέργειας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αλλά και για την τροφοδοσία μετά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Εάν φορτίζονται οι μπαταρίες με ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται από εργοστάσια που καίνε κάρβουνο, αντιλαμβάνεστε τότε βέβαια ότι ο στόχος της σημείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος δεν εξυπηρετείται. Έτσι λοιπόν πρέπει να εξεταστεί ολόκληρη αυτή η αλυσίδα, όχι μονάχα το τμήμα αυτοκίνητο αλλά και η παραγωγή του. Πώς είναι η κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή των αυτοκινήτων. Οι ε, αυτοκινητοβιομηχανίες ακολουθούν μια καινοτομία και για την παραγωγή του αυτοκινήτου. Αυτά όλα πρέπει να περιληφθούν στην νέα νομοθεσία. κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί, κύριε Ούλμερ, η έκθεσή σας τον Ιούνιο, έκτο δηλαδή στην Ολομέλεια. Φτάνουμε τώρα στο τέλος της ημερησίας διατάξεως. Ευχαριστώ λοιπόν και επισημένο ότι, χωρίς να φταίμε θα έλεγα, αλλά με την ανάληψη καθηκόντων του νέου Πάπα, αναγκάζεται να γίνει σήμερα η ανοιχτή διάσκεψη των Προέδρων. Αποφάσισα λοιπόν ότι θα αναβάλουμε την έναρξη συνεδριάσεώ μα μέχρι τι 4 παρατέταρτο, ώστε όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανοιχτή αυτή διάσκεψη των Προέδρων να μπορέσουν να δουν τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Αλλά έχουμε και άλλε σημαντικέ εκθέσει σήμερα και έτσι λοιπόν παρακαλώ όλοι και όλε να είστε παρούσε και παρόντε στι 4 παρατέταρτο. Θα γίνει πρώτα ψηφοφορία και αμέσω μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση τη ε, ε, εκθέσεω τη κυρία Γκλένη Βίλκοτ. Έχουμε και προσκεκλημένο σήμερα μαζί μας τον κύριο Ταϊάννη για θέματα αυτοκινήτου πάλι. Θα είναι είδος παιχνιδιού πινκ-πονκ το απόγευμα με ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα γίνει συζήτηση, θα μπορέσουμε να θέσουμε τις απαραίτητες ερωτήσεις και να λάβουμε τις απαραίτητες απαντήσεις όλοι είστε προσκεκλημένε και προσκεκλημένοι να συμμετάσχετε στη συζήτηση και εσείς όσοι κάθεστε στις πίσω, στα πίσω, πίσω θέσεις και από τις 18 και 30 μέχρι τις 19 και 15 θα συζητηθεί 18 και 30 έως 19 και 15, δηλαδή 45 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας για την έκθεση. Παρακαλώ, ο σχεδιασμός σας να είναι τέτοιος και για τους ε, συναδέλφους βουλευτές και για τους συνεργάτες ε, ώστε να ανταποκριθείτε στην ε, πρόβλεψη αυτή. Σας εύχομαι καλό μεσημεριανό διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε στις 4 πάντα.